Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. <coughs> Καθίστε παρακάτω. Για να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας σήμερα το πρωί. Είναι η δεύτερη μέρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Ρέντζι. Πρώτο σημείο στην ημέρησια διάταξη είναι η έκθεση πρωτοβουλία για τους ε, θεματικούς στόχους σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η έκθεση αυτή εστιάζει στις κύριες προκλήσεις για να επιτύχουμε την υλοποίηση των θεματικών στόχων και προχωρεί και σε μια ανάλυση <clears throat> των συνεργειών που επιτρέπουν μια καλύτερη υλοποίηση. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης μια αξιολόγηση του πώς η υλοποίηση των θεματικών στόχων έχει εξασφαλίσει να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες στον τομέα των επενδύσεων και υποστηρίζει τη λειτουργικότητα, λειτουργικότητα σε επενδύσεις αυτές. Το Νοέμβριο η συγγήτριά μας παρουσίασε αρχικές της θέσεις και τώρα παρουσιάζει το σχέδιο έκθεσης της αν <clears throat> προθεσμία ε, κατάθεση τροπολογιών είναι το μεσημέρι της 25ης Φεβρουαρίου ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Απρίλιο. Μέχρι τις 10 έχουμε χρόνο να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Εάν χρειαστεί θα πρέπει να περιορίσω το χρόνο αγόρευσης και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι πήραμε σήμερα μια ενημέρωση από το Τμήμα Έρευνας και σας ευχαριστώ που το δώσατε εγκαίρως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για το Λοιπόν, κύριε Μάτ, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που <clears throat> έχουν συμφωνήσει να συζητήσουμε το τόσο σημαντικό θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τους κοιόδες συζητητές πρέπει να πω εξ αρχής ότι είχαν καταδείξει ένα πνεύμα συνεργασίας ένα πολύ θετικό πνεύμα. Η έκθεση αυτή λοιπόν αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι προφανώς σημαντικές για την οικονομία των ευρωπαϊκών περιφερειών και για την απασχόληση και για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδίω έχουν μια μεγάλη ευθύνη για τα θέματα αυτά, ιδίω σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χρονικό διάστημα 2014-2020 ε, έχουν δοθεί 27 εκατομμύρια ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας <clears throat> και να μπορέσουν να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό περιλαμβάνει συνεργατικές επιχειρήσεις και κοινωνικού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Ο στόχος 3 του οποίου ανα, ανατέμνεται η εφαρμογή σε αυτή την έκθεση έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί έχει εστιάσει στην πρόθεση του επιχειρήν, στην πρόθεση και την υλοποίηση νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας και δημιουργία νέων υπηρεσιών για να υποστηρίξουν την ε, ανάπτυξη αγορών σε εθνικό αλλά και κυρίως σε διεθνές επίπεδο. Υπήρξε μια σημαντική ε, ποσόστοση για 94 δισεκατομμύρια μαζί με τις εθνικές συνεισφορές. Το Κοινοβούλιο όμως έχει υπογραμμίσει πάντα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο, <clears throat> η σπονδυλική στήλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτή η ίδια αντίληψη διατρέχει όλη την έκθεσή μου που αντιμετωπίζει διάφορα εγκάσια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το τονίσουμε ιδιαίτερα. Αναφέρομαι σε όλες αυτές τις πτυχές και τα προβλήματα που εμποδίζουν την βιώσιμη και αποτελεσματική εφαρμογή των επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η απλοποίηση λοιπόν και η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία που έχουμε για να προωθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών και αρχών. Είναι πολύ σημαντικά σημεία τα οποία θίγουμε εδώ. Ένα άλλο θέμα ουσιαστικό είναι η αρχή της εταιρικής σχέσης, που συχνά ε, εφαρμόζεται μόνο τυπικά και εις βάρος πολλών άλλων οικονομικών και κοινωνικών φορέων. Όμως ε, που είναι πολύ καλά εγκατεστημένοι σε τοπικό επίπεδο και γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες της περιοχής. Ήθελα επίσης ε, σε αυτή την δύσκολη περίοδο να πω και κάτι άλλο. Μιλάω για την διασύνδεση της, ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το μεταναστευτικό πρόβλημα. Συχνά, ε, επειδή βρίσκονται ακριβώς σε περιοχές όπου ε, υποδέχονται τους μετανάστες, παίζουν σημαντικό ρόλο. Επίσης παίζουν καινοτόμο ρόλο ακόμα και μέσα σε παραδοσιακά σχήματα. Επίσης, το θέμα της ε, κυκλικής οικονομίας μπορεί να βοηθήσει σε μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης ποιοτικέ, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις της COP21 στο Παρίσι. Και τα δύο αυτά σημεία θα μπορούσαν να ενταχθούν στον θεματικό στόχο 3, ούτως ώστε στις, ε, στο μέλλον να ληφθούν υπόψη αυτά τα βήματα προς τα εμπρός και θα έχουν επιπτώσεις και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό η Ευρώπη δεν πρέπει να μείνει πίσω. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Ε, το σχέδιο της έκθεσης είναι στη διάθεσή σας. Επομένως, περιμένω και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία μεταξύ, ε, μεταξύ μας, όπως είχαμε και μέχρι τώρα, για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Τσίκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Νταμάτο. Η έκθεσή της συνολικά είναι θετική. Είναι πλούσια με στοιχεία τα οποία αξίζει να μας απασχολήσουν. Φυσικά, πριν φτάσουμε εδώ, έγινε μια ενδελεχής ανταλλαγή απόψεων, έγινε μια αντιπαράθεση απόψεων και με, τις, ε, με την τοποθέτηση και την ε, σύγκριση των ιδεών ανάμεσα στην κυρία Μάτο και στους σκιώδεις ηγητές. Εγώ εκπροσωπώ και τον συντονιστή, τον κύριο Βανίστερ Ρόι και κάποιους άλλους συναδέλφους. Στην έκθεση 4 της έκθεσης, κατά τη γνώμη μου, με βάση τα όσα μου είπαν και οι συνάδελφοι, ε, γίνεται μια πολύ μικρή αναφορά στην πρόσβαση στην πίστοση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολύ ανεπαρκής. Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και προτεραιότητα. και θα προτιμούσα να έχουμε μία παράγραφο ολόκληρη για το θέμα αυτό και να ζητήσουμε με έμφαση να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ μέσω της πραγματικής, μια μιας επαρκούς ροής χρήματος. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υποφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, λόγω της συγκυριακής κρίσης αυτής. Όλες οι διαδικασίες που στο, στόχο έχουν να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις, οι διαγωνισμοί κτλ. Ε, είναι, γίνονται ε, συχνά εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων. Ε, συχνά ε, δεν λαμβάνουν ε, τις ανακοινώσεις για την υποβολή προσφορών, ας πούμε, εγκαίρως. βρίσκουν το 30% της χρηματοδότησης εν γέννη, αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία, το 70% λείπει. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το θέμα της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σε ό,τι αφορά την, το βάλτομα που έχουν οι εσωτερική, εσωτερική αγορά ε, δεδομένης της κρίσης είναι πολύ πιο σημαντικό να έχουν διέξοδο, να έχουν ε, ε, καλά στελέχη, να ανοίξουν προς το εξωτερικό. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ε, χρησιμεύουν για την ανάπτυξή τους. Νομίζω ότι αυτή η ιδέα της διεθνοποίησης πρέπει να αξιοποιηθεί. Μόνο 25% το ΜΜΕ ε, λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο και το 13% μόνο πραγματικά δραστηριοποιείται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε αυτό που είπα έλεγα πριν. Άμεσες και έμεσες, ε, άμεσα και έμεσα κονδύλια. Γιατί σήμερα οι ΜΜΕ ε, έχουν πάρα πολλές δυσκολίες για να βρουν τη συγχρηματοδότηση που χρειάζεται για να συμμετάσχουν σε διάφορα προγράμματα. Θα τόνιζα λοιπόν πάρα πολύ το θέμα της εισρωής ε, κεφαλαίων και θα ήθελα ε, αυτό να αναφερθεί με μεγαλύτερη έμφαση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Yes, Mr. Uh, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη συνάδελφο Ταμάτο για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της νομοδότησής της. Της έκθεσης. Συμφωνώ απολύτως με τη δήλωση ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το καιρό έχουμε διαπραγματεύσεις για ε, μια συμφωνία ή περισσότερες συμφωνίες ε, ελευθέρων συναλλαγών και πρέπει να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες μας για να μπορέσουν να σταθούν σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά με τέτοιο ανταγωνισμό. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι ήδη από το προσχέδιο της νομοδότησής της η κυρία Νταμάτο αναφέρει την κυκλική οικονομία και τη θεωρεί βάση για οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη ε, της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες. Διότι ε, εκεί οι μικρομεσαίες δημιουργούν θέσεις απασχόλησης στην ε, παραδοσιακή οικονομία, αλλά στην κυκλική οικονομία χρειαζόμαστε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ε, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση συσκευών, επισκευές. Αυτά είναι κάποια επαγγέλματα που σχεδόν έχουν χαθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Έχουν εγκαταληφθεί και θα πρέπει να τα ξαναβρούμε. Βεβαίω, οι μικρομεσαίες μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας κάθε φορά, γι' αυτό και καλούμεθα να εξαντλήσουμε το δυναμικό και τις δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας. Θέλω να τονίσω κάτι ακόμα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται οπωσδήποτε εύκολη πρόσβαση ε, σε κεφάλαια και θα πρέπει να διευκολύνονται για το σκοπό αυτό. Ιδιαίτερα για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Διαρθρωτικά και Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, αλλά και για τις εμπορικές τράπεζες. Θα πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν μια πλατφόρμα για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών για να δούμε πώς στηρίχθηκαν οι μικρομεσαίες την τελευταία προγραμματική περίοδο. Και αυτές οι μέθοδοι που έχουν επιτύχει στην πράξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθηθούν νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοφυείς, για να σταθούν στα πόδια τους και να βγουν στην αγορά. Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να τονιστεί μάλλον περισσότερο στην ομοδότηση είναι το εξή. Πρέπει να σταματήσει αυτή η Αναντιστοιχεία που υπάρχει ανάμεσα στην παιδεία και στην οικονομία. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να έχει και μάθημα για το επιχειρήν. Πώς μπορεί κανείς να ιδρύσει μια επιχείρηση, να τη λειτουργεί με επιτυχία και να μπορεί να ε, χρησιμοποιεί και τις οικονομικές δυνατότητες που ανοίγονται μεταξύ αυτών και ε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα διευθυντικά ταμεία. Και για τις στατιστικές πρέπει να πω ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις επιχειρήσεις και θα πρέπει να τονιστεί και αυτό στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Να φροντίσουμε να υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο και στο επιχειρηματικό γίγνεσθε. Για να συμβεί αυτό βέβαια πρέπει να πέσουν ακόμα πολλά εμπόδια και φραγμοί που στέκουν και εμποδίζουν τις γυναίκες να δραστηριοποιηθούν ως επιχειρηματίες και οικονομικά εμπόδια. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόεδρος ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάκοφτσιτς, εξ ονόματος του κυρίου Στροβίτσιους, που είναι σκιώδης. Ε, ευχαριστώ. Ο σκιώδης ηγητής κ. Στρεβίτσιος απουσιάζει και θα μιλήσω εξ ονόματός του αλλά και εξ ονόματος της σύνολης ομάδας των φιλελευθέρων. Η κυρία Ανταμάτο ήδη πρέπει να πω έχει κάνει μια εξαιρετική γνωμοδότηση. Επιτρέψτε μου να προσθέσω και εγώ μερικά λόγια από πλευρά των φιλελευθέρων. Το πρώτο έχει να κάνει με τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη λεγόμενη ψηφιακή εποχή. Νομίζω ότι αυτό δεν το τονίζει αρκετά η γνωμοδότηση. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη σημασία συμμετοχή των μικρομεσαίων σε όλες τις τεχνολογικές και ψηφιακές εξελίξεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εδώ καλών και βελτίστων πρακτικών. Θα ήθελα όμως να καλέσω την εισηγήτρια να το λάβει υπόψη της, να το συνειδητοποιήσει περισσότερο και να καταλάβει και αυτά τα νέα φαινόμενα στη ψηφιακή εποχή που έχουν τεράστια σημασία και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και θα ήθελα να το δω και στη γνωμοδότηση αυτό. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με του ΣΟΤΑ και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Εμείς είμαστε Επιτροπή περιφερικής ανάπτυξης. Και ε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει και πώς μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις μικρομεσαίες πόλεις, για παράδειγμα. Αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και την αστική και την ανάπτυξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Επίσης, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ή ακόμα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό. Υπάρχουν ήδη τέτοια δίκτυα, αλλά πρέπει να τονίσουμε τις μικρομεσαίες. Α, έφτασε ο κύριος Στρεβίσιους, ο σκιώδης ηγητής μας, ε, στο μεταξύ, αλλά νομίζω ότι τον κάλυψα και εκείνον με τα λεγόμενά μου. Sorry, Mr. has oh, <laughs> <laughs> Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πράγματι. Θα μπορούσα να σας προσφέρω μια κάσα σαμπάνιας και κόκκινου και άσπρου κρασιού από την Κροατία που είναι εξαιρετικής ποιότητας, όλα αυτά για την περιφερειακή ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ που ξεκίνησα την παρουσίαση για το σχέδιο έκθεσης περί της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων και χαίρομαι πάρα πολύ για τις ε, προσπάθειες των σκιωδών εισηγητών και του εισηγητή και τη συνεργασία που είχαμε. Άκουσε ο εισηγητή όλα τα επιχειρηματά μα. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Υπάρχουν ορισμένε πτυχέ όμω οι οποίε θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν <clears throat> πιο εντατικά. Αυτό είναι μια φυσιολογική διαδικασία για την βελτίωση τη έκθεση αυτή. και με την αδειά σας θα αναφέρω ορισμένα από αυτά τα θέματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω εστίασης και να σα δώσω επίσης και κάποια σκέψεις για το τι θα μπορούσε να περιληφθεί στις τροπολογίες μας. Παραδείγματο χάρη, όταν ζητούμε καλύτερη συνεργασία και συνεκτικότητα μεταξύ των πολιτικών επενδύσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπω πρέπει να αναφέρουμε και την Ένωση Αγορών, <clears throat> που είναι σημαντικό στοιχείο του σχεδίου επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη και για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε ένα σαφή δρόμο <clears throat> για την αξιοποίηση όλων των κεφαλαιοχικών πόρων για όλες τις μικρομεσαίες επιχείρησεις. Ένα θέμα το οποίο υπογραμμίζουμε συνέχεια. Εναλλακτικέ και πιο διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης <clears throat> και άρση περιττών φραγμών εξακολουθούν να υπάρχουν αυτοί οι φραγμοί ακόμα για τις διαμεθοριακές επενδύσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις επενδύσεις και, και το επιχειρήν και για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για το επιχειρήν και για τις επενδύσεις. Επίσης, για τις ψηφιακές δεξιότητες. Αλλάζει το ψηφιακό τοπίο. Η αγορά εργασίας τροποποιείται δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες. Ας είμαστε ειλικρινείς για το θέμα αυτό. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν πρωτοβουλίε για να υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση στο ψηφιακό τμήμα της παιδείας, ώστε η παιδεία να είναι πραγματικά προσαρμοσμένη στις αναπτυσσόμενες αγορές που χρειάζεται η βιομηχανία, αγορές εργασίας και επίσης θα πρέπει να δώσουμε την κατάλληλη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση για τους εργαζόμενους και τους ετούντες εργασίας ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την πρόοδο την, <clears throat> στο τεχνολογικό τμήμα της αγοράς. Τρίτον, για ό,τι αφορά τις κοινωνικές επιχείρησεις που είναι κέρυες για την κοινωνική καινοτομία και οι οποίες επίσης <clears throat> ασκούν ένα μεγάλο αριθμό από εμπορικές δραστηριότητες. Είναι απαραίτητο να έχουμε υπόψη μας ότι δίνουν πάρα πολλά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή ενία Αγορά και δημιουργούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, μεταλαμπάδευση γνώσεων σε σχέση με αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Και επίσης να δημιουργήσουμε κέντρα για αυτές τις επιχειρήσεις, κέντρα εκόλαψης και επιτάχυνσης της δημιουργίας <clears throat> τέτοιων επιχειρήσεων. Θέλω να τονίσω επίση και το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ακόμα και αν αυτό αναφέρεται στην, ε, στο σχέδιο έκθεσης, ακούγοντας αυτά που λένε οι εκλεγμένοι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θεωρούν ότι δεν έχουν εμπλακεί επαρκώς στην ε, διαμόρφωση της πολιτικής για τα θέματα αυτά. Ο ρόλος ο οποίος τους αποδίδεται πολλές φορές είναι <clears throat> όχι εταίρου, αλλά απλώ εμπλεκομένου σε δευτερεύον επίπεδο. Για να μπορέσουμε θα πρέπει, για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να εμπλέξουμε πολύ περισσότερο και πολύ πιο έγκυρα τους τοπικούς και περιφερειακούς ε, εκλεγμένους. Πιστεύω ότι με όλες αυτές τις προτάσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, ώστε η έκθεση μας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να είναι πιο επωφέλης. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που ήρθε εγκαίρος ο σκιώδη εισηγητής και μπόρεσε να συμμετάσχει. Κυρία Τόμασιτς, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Νταμάτο για τη θαυμάσια έκθεση, για την αποτελεσματική συνεργασία και το αποτέλεσμα είναι μια καλά διατυπωμένη έκθεση. Εμείς υποστηρίζουμε το σχέδιο έκθεσης, αλλά θα ήθελα να προσθέσουμε κάποια στοιχεία που αφορούν τα βασικά προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διοικητικό άχθος, ε, περιπλοκότητα των συστημάτων ενίσχυσης, ε, νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις. Πιστεύουμε ότι τα προβλήματα θα μπορούσαν να επιληθούν με την συμπερίληψη της πολιτικής συνοχής στην πρωτοβουλία για το ευνομοθετήν, ε, καλύτερη διασύνδεση των ταμείων, δημιουργία δυναμικού των τοπικών αρχών κοινέ καταρτήσεις μεταξύ των τοπικών αρχών και των ε, stakeholders, κοινά προγράμματα για τις αρχές διαχείρισης και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, προσπάθεια να, τους, να τις βοηθήσουμε, το coaching και βοήθεια για την ε, εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη συμμετοχή στα προγράμματα. Ο σκιώδης συγητής ο κ. Κουτσολίνο, πολύ σύντομα. Και εγώ έχω θετική γνώμη από τη συνεργασία που είχαμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Νομίζω ότι τελικά θα μπορέσουμε να έχουμε μία έκθεση ισορροπημένη, η οποία θα διατηρήσει έτσι, μία στρατηγική θεώρηση ε, εστίασης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά θα θέσει επίσης ε, και άλλα θέματα και ερωτηματικά, κυρίως που αφορούν τα διάφορα συστήματα ενίσχυσης που υπάρχουν προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των διαρθωτικών ταμείων. Κυρίως τα θέματα της πίστοσης από τις ε, τράπεζες. Πρέπει να δοθεί εκεί μεγαλύτερη έμφαση. Είναι λεπτό το θέμα, είναι το, το θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης. Πώς θα μπορέσει αυτή η διακυβέρνηση να είναι πιο διαφανής, πιο αποτελεσματική σε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι να χρηματοδοτεί επιλεκτικά ή με το σταγονόμετρο ή να αφήνει ας πούμε δημόσιους πόρους σε αγρανάπαυση. Δεν γίνονται αυτά. Ε, νομίζω ότι η έκθεση τα θέτει αυτά τα θέματα. Μία παρατηρήση, τα, τα ξέρει αυτά η κυρία Νταμάτο. Όχι μόνο τα σημεία στα οποία στέκεται εκείνη στην έκθεσή της, δηλαδή τα βασικά ε, περιβαλλοντικά θέματα, τις ε, βασικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλά το θέμα, βασικό θέμα της κοινωνικής καινοτομία. Το είπα και θα το ξαναπώ. Νομίζω ότι μπορούμε τις επόμενες ώρες κάτι να σκεφτούμε γύρω από αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Μια μοντέρνα ε, ανταγωνιστική επιχείρηση τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη χρειάζεται να θέσει έμφαση όχι μόνο σε μεγάλες προκλήσεις που συνδέονται με μια πιο βιώσιμη οικονομία που θα συνδέεται περισσότερο και θα λαμβάνει υπόψη τα, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις τα επόμενα χρόνια, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θέμα της κοινωνικής καινοτομίας. Είναι σημαντικό αυτό για την νέα επιχείρηση τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια παρατήρηση πάνω σε αυτό, να, να βρούμε τη διατύπωση, την κατάσταση στις επόμενες ώρες, αλλά γενικά έχω θετική γνώμη για την έκθεση συνταμάτων. κύριος Ρόπε. Ευχαριστώ. Σήμερα είναι η 16η Φεβρουαρίου και η Λιθουανία ε, υπάρχει ως κράτος επί 98 χρόνια. Είναι η επέτειος της ίδρυσης του κράτους μας. Συζητάμε πολύ σημαντικά θέματα σήμερα. και θα μπορούσαμε, ε, αν λύσουμε το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να εξασφαλίσουμε περισσότερε θέσει απασχόληση και έσοδα για την Ευρώπη. Χαίρομαι που έθεσε η συγκήτρια αυτά τα θέματα. Όταν μιλάμε για τι μικρομεσαίε, όλοι συμφωνούμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά τη ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι η λύση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τη ανεργία. Θα πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν σε αυτά τα ταμεία και να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τα ποσά των ταμείων αυτών το ποσοστό απορρόφησης διαφέρει από κράτος σε κράτος, αλλά πολλά κράτη-μέλη ε, καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν 100% τα κονδύλια που τους ε, προσφέρονται. Είναι σημαντικό επίσης να εμπλέξουμε και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε αυτή την προσπάθεια. Διάφορα προγράμματα εφαρμόζονται στις πόλεις, βέβαια, αλλά είναι σημαντικό αυτά τα προγράμματα να εξαπλωθούν σε, σε, μια, σε όλες τις περιφέρειες, όχι μόνο στις πόλεις. Αυτά τα προγράμματα επίσης είναι σημαντικά για τη φορολογία σε πολλά κράτη-μέλη, για την, τα φορολογικά έσοδα. Παραδείγματος χάρη, μια τεχνολογική εταιρεία, η οποία αποφεύγει να πληρώσει α, φόρους. Υπάρχουν τέτοιες εταιρείες που φοροδιαφεύγουν με ποσά ύψους, ας πούμε, ενός δις. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα μεταξύ διαφόρων ευρωπαϊκών εταιρείων, αλλά και ευρωπαϊκών και ξένων. Ούτως ώστε οι εταιρείε αυτές να δραστηριοποιούνται και να δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Ευχαριστώ κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έκθεση, να την καλωσορίσω και να ευχαριστήσω την συντάκτρια της νομοδότησης, κυρία Νταμάτο. Τονίζεται πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως είναι η μείωση του γραφειοκρατικού άχθους, ε, επιτάχυση της υλοποίησης, διάδοση της γνώσης στα κράτη-μέλη και άλλα τεινά απευθυντική θηρίδα, αυτό το one-stop shop ε, σε περιφερειακό επίπεδο για ενημέρωση έως προ την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και επίσης τονίζεται την ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρμογή όλων αυτών. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε, να σκεφτούμε την αρχή της εταιρικής σχέσης και της ε, ε, διάδοση αυτής της αρχής θα πρέπει να εισαχθεί, να γίνει κτήμα και να διαδοθεί. Όχι μόνο από το στάδιο της χάραξης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των ΕΣΠΑ, αλλά όταν και προκυρήσουμε, ε, και όταν προκυρήσουμε διαγωνισμούς για την υποβολή έργων και ε, εκδήλωση ενδιαφέροντος, διότι στα κράτη-μέλη έχουν ε, υπάρξει περιπτώσει ε, που προκυρήσουν διαγωνισμούς ανοιχτούς και μετά από ένα χρόνο έχουν υπογράψει τις εξής συμβάσεις αριθμός 2. Ε, δηλαδή κάτι τρέχει με τους διαγωνισμούς, με τα κριτήρια, με τον τρόπο υποβολής που δεν ε, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες τους. Σήμερα χρειάζονται χρηματοδότηση, όχι δάνεια, κυρίως επιδοτήσεις και δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν, γιατί δεν γνωρίζουν καλά τα κριτήρια ή δεν έχει σχεδιαστεί καλά ο διαγωνισμός και η προκήρυξη. Αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να ε, φροντίζουν να πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους. Και ένα άλλο πρόβλημα που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στην πράξη είναι ότι υπάρχει θέμα χρηματοδότησης και πρόσβασης αυτή. και ε, επηρεάζει πάρα πολύ η πιστοληπτική ικανότητα μιας χώρας ε, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, γιατί μπορεί οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μετά υπάρχει και το σκέλος της συνυπευθυνότητας της συγχρηματοδότηση από τον κρατικό προπολογισμό που χωλαίνει. Το συζητήσαμε και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, μάλλον πρέπει να το συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Κύριος Έθριτζ. Ευχαριστώ. <clears throat> Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η συζήτηση γιατί πρωτού εκλεγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήμουν ενεργός στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είχα μια δική μου επιχείρηση εδώ και πολύ καιρό. Το διάστημα αυτό, αυτό το οποίο με περισσότερο ήταν πιο χαμηλή και πιο απλή φορολόγηση, λιγότερο χαρτοβασίλειο καλύτερη πρόσβαση σε εκπαιδευμένους εργαζόμενους και λιγότερη φραγμή στο διεθνές εμπόριο, αγορά και πώληση προϊόντων. <clears throat> και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει υποθέτω και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο δεν με ενδιαφέρε ούτε εμένα ούτε τους συναδέλφους μου ήταν η κοινωνική καινοτομία, η βιωσιμότητα και το περιβάλλον. Γιατί λεφτά προσπαθούσαμε να βγάλουμε προσπαθούσαμε να βγάλουμε λεφτά και να απασχολούμε ανθρώπους. Πιστεύω ότι αν έχουμε τις σωστές προϋποθέσεις σε μια χώρα, <clears throat> μπορείτε να έχετε μια καλή επιχείρηση η οποία θα προσελκύσει επενδύσεις. Δεν χρειάζεστε πάντα να έχετε τις κυβερνήσεις να επενδύουν για να γίνει κάτι. Είναι ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή, θα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση και προσβλέπω σε αυτήν, αλλά από την πλευρά κάποιου ο οποίος έχει πράγματι δουλέψει σε μικρομεσαίες επιχείρησεις, ας προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στη λιγότερη ρύθμιση, στο λιγότερο χαρτοβασίλειο και να εστιάσουμε σε αυτούς οι οποίοι δημιουργούν πλούτο και επομένως δημιουργούν τα δαπανίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ο κύριος Φαν Νίστλεροι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ πάρα πολύ για την γνωμοδότηση και για το χρόνο ε, στον οποίο ήρθε την εισηγήτρια Μπράβο σας. Πολύ Πολύ πρόσφατη ήταν η συζήτηση που είχαμε ε, για ε, την εφαρμογή. Ήταν η έκθεση Βεζιά και τώρα πάρα πολύ γρήγορα έχει φέρει τη γνωμοδότηση. Πολύ καλό παράδειγμα προς μίμηση για το πώς μπορεί κανείς να δραστηριοποιείται και να επηρεάζει σημαντικά στοιχεία της περιφερειακής πολιτικής. Μερικά σχόλια έχω. Ε, Πρώτον, Κοιτάει τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών η συγκήτρια. Αν δούμε στην εφαρμογή τι γίνεται, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν χώρες που τα πηγαίνουν πολύ καλά. Το γράφει και στην αιτιολογική έκθεση. Για ποιο λόγο ε, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν τόσο καλές επιδόσεις και άλλα όχι. Σήμερα πήραμε τη νέα έρευνα ε, που έγινε ε, για την έκθεσή σας και λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Ποια είναι αυτά τα κράτη-μέλη. Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Βουλγαρία, Ρουμανία, τα πάνε πολύ καλά, Φιλανδία. Βέβαια, όταν πρόκειται για πρωτοβολίες στο μικρομεσαίων και κάπου αλλού λέει τώρα ε, για άλλες χώρες που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην έκθεση εφαρμογής ε, εγώ αναρωτιέμαι πώς είναι των πέντε χώρες να τα πηγαίνουν τόσο καλά ενώ κάποιες άλλες υπολείπονται και χωλένουν. Έχω κανονική εικόνα ή στρεβλή, να μου το πείτε, με ενδιαφέρει. Επίσης, με έχουν εντυπωσιάσει και τα αριθμητικά στοιχεία στο, στο άρθρο 16.3. 94 δις παρακαλώ είναι το συνολικό ποσό, 94 εκατομμύρια στην τρέχουσα περίοδο. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Στη συζήτηση ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη συνοχή και για τα κονδύλια και τα ταμεία μας, είναι πολλά τα λεφτά. <laughs> Ε, αν βλέπουμε τη συζήτηση στην Ήτρε, στην Επιτροπή Βιομηχανίας για τις Μικρομεσαίες, μιλάμε για μέσα βοήθειας, χρηματοδότησης και ξέρουμε ότι υπάρχουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις όμως από τη δική μας σκοπιά είναι το διπλό, το διπλάσιο σε σχέση με την περασμένη προγραμματική περίοδο και ε, η θεματική συγκέντρωση είναι προτεραιότητα. Ε, και βάσει ε, αυτή συντάχθηκε και ο νέος κανονισμός για την, ένα, για τη νέα προγραμματική περίοδο. Και στο σημείο 3 ε, αναφέρεται η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι τόσο σπουδαίο το αποτέλεσμα, αλλά θα πρέπει να προβάλλεται κιόλα και να το γνωρίζει ο κόσμος. Και με καθησυχάζει αυτό που βλέπω ότι ε, γίνονται επενδύσεις και θα πηγαίνουν καλά κάποιες χώρες. Ε, στο συγκεκριμένο έγγραφο γίνονται και κάποιες συστάσεις από την υπηρεσίες αλλά και από την Επιτροπή των Περιφερειών από ανεξάρτητες ερευνητικές υπηρεσίες και γίνεται λόγος για συνέργειες. Και κάτι μου λείπει εκεί. Εσείς το λέτε βέβαια στη γνωμοδότησή σας, στην αιτιολογική έκθεση, στη δική μου σελίδα 9 συγκεκριμένα, αλλά αν κοιτάξετε Πώς μπορεί κάποιος μικρομεσαίος να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου ή κεφάλαια γενικότερα. Αυτόν δεν τον νοιάζει πάρα πολύ αν θα προέρχεται από τα διορθωτικά ταμεία ή από το ΕΦΣΙ, από εγγυήσει, από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή από που θα έρθουν. Γιατί έχουμε και αυτό το καινούριο φιντάνι τώρα, το ΕΦΣΙ. Αυτό που θέλει ο επιχειρηματίας είναι ε, Πώ θα τα μάθει όλα αυτά, να μην έχει εκατοθυρίδε που θα πρέπει να τρέχει να ενημερώνεται, αλλά να τα ξέρει γρήγορα και εύκολα. Και αυτό με τις συνέργειες νομίζω δεν έχει καλυφθεί πάρα πολύ στη γνωμοδότηση. Θα πρέπει να κοιτάξουμε ποια είναι η δικιά μας θέση στα συνολικά εργαλεία και μέσα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε πώς θα τα εφαρμόσουμε. Και αν εμείς ε, διευκολύνουμε τα πράγματα ή όχι. Αυτά. Και μια τελευταία παρατήρηση Τώρα αυτό τον καιρό τρέχει μια πρωτοβουλία για να ενισχυθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι startups. Ε, είναι πάρα πολλές αυτές οι εταιρείε που ψάχνουν μια ευκαιρία να ε, μεταφράσουν μια ιδέα που έχουν στην πράξη. Τώρα, όταν είσαι startup, πώς θα γίνεις κανονική επιχείρηση. Αυτό είναι το θέμα και τι δυνατότητες θα έχεις και τι ευκαιρίες. Οι μικροπιστώσεις δίνονται πιο εύκολα για ε, πολύ μικρά ποσά. Είναι και άλλοι τρόποι καινούργοι, το crowdfunding κλπ. Αλλά αυτή τη στιγμή ε, φεύγεις από τάξη μεγέθους 1-2 εκατομμύρια και φτάνεις στα 100 εκατομμύρια, οι τράπεζες κάπως διστάζουν να σε χρηματοδοτήσουν. Ε, αυτό είναι λοιπόν πώς θα γίνει το βήμα από τη νεοφυή επιχείρηση να γίνει μια μικρομεσαία. Σα ερωτώ και πάλι λοιπόν, γιατί κάποιες χώρες έχουν καλές επιδόσεις και κάποιες άλλες όχι. Δεύτερον, τι γίνεται με τις συνέργειε και τρίτον, τι γίνεται με τις startups. Και θα μας πείτε, αν έχετε λάβει υπόψη αυτή τη μελέτη ε, που έχει σχέση και με τη δική σας νομοδότηση. Αλλιώ να κάνουμε τροπολογίες εμείς από την πλευρά μας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριος Κόλιν Γουλφ και ο κύριος Μάρεκ Πρέζορ. Ποιο θα πάρει το λόγο, τους δυο σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι τμήματάρχης ε, ε, στην ε, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης Άκουσα με μεγάλη προσοχή τη συζήτηση και διάβασα επίσης πολύ προσεκτικά την έκθεση. Στη συζήτηση ακούστηκε, ακούστηκαν σχόλια για τη σημασία ε, βελτίωσης των οικονομικών ροών, της, της οικονομικής χρηματοδότησης. Πιο εύκολη πρόσβαση σε εναλλακτικέ πηγές χρηματοδότησης. Απλούστευση επίσης των διαδικασιών και θα πρέπει οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης να μπουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Ε, δημιουργία δυναμικού, βελτίωση της διακυβέρνησης, ε, βελτίωση της διαφάνειας, εμπλοκή των διαφόρων φορέων, ε, καλύτερες εταιρικέ σχέσεις και καλύτερη χρησιμοποίηση των ε, ειδημόνων στις περιφέρειες και κυρίως στις πόλεις, ούτως ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. συνεργασία για την ε, μείωση των φραγμών στο εμπόδιο, διεθνοποίηση, συνεργασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατέγραψα τις μεγαλύτερες δυνατότητες για μεγαλύτερη έρευνα και ανάλυση στο γιατί κάπου λειτουργούν τα πράγματα καλύτερα και για και τι μπορούμε να κάνουμε αλλού για να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες ε, πλατφόρμες για διάδοση των καλών πρακτικών και καλών προσεγγίσεων. Για την ουσία τώρα της δουλειάς, σημαντικό είναι ότι δίνεται έμφαση στη βελτίωση των ε, δεξιοτήτων και της κοινωνικής ε, οικονομίας και των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας. Το τι κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα επιχειρησιακά προγράμματα εστιάσουν καλύτερα τώρα στις στρατηγικές προτεραιότητες και κυρίως στο να εξασφαλίσουν ότι η υποστήριξη για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις όντως δίδεται. Τα προγράμματα επιλέγονται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Ε, δίνουμε ε, μεγαλύτερη έμφαση ε, στις τεχνολογικές επιχειρήσεις, δημιουργία value chains, ξυγχρονισμός των ε, εργασιών, υποστήριξη δεξιοτήτων, μεγαλύτερη έμφαση στο να δοθούν επίσης αυτές οι πλατφόρμες υποστήριξης και δικτύωσης, ε, μεταφορά της τεχνολογικής γνώσης και αναβάθμιση των μηχανισμών, ούτως ώστε να υποστηρίξουμε τις νεοφύης επιχειρήσεις, επιχειρήσεις και να μπορέσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω. Ε, Αναφέρθηκε επίσης ε, το άρθρο 16. 800.000 ε, περίπου επιχειρήσεις αναφέρεται ότι θα επωφεληθούν από την υποστήριξη αυτή την περίοδο και 140.000 ε, είναι νεοφύης επιχειρήσεις από τις 800.000. Επίσης, για την υποστήριξη ελπίζουμε ότι περίπου η μισή υποστήριξη θα περάσει μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και προσπαθούμε να τελεσφορήσει αυτή τη διαδικασία όσο γίνεται. Τώρα κάποια συγκεκριμένα σημεία σε σχέση με την απλούστευση. Δουλεύουμε εργοδός ούτως ώστε να υλοποιήσουμε αυτά που συστήνει η ομάδα υψηλού επίπεδου για τη μείωση του διοικητικού άχθους ε, για τους δικαιούχους και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ε, ΜΜΕ. Για τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης που θα πρέπει να είναι στο ίδιο πλαίσιο για να υπάρχει μια συνέργεια. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα εργαλεία λειτουργούν, ε, κυρίως του ορίζοντα 2020 και τα ευρωπαϊκά διαρθωτικά και επενδυτικά ταμεία, ε, προσέγγιση για, για την αριστεία, προγράμματα τα οποία έχουν περάσει τη διαδικασία επιλογής σε σχέση με τον ορίζοντα 2020, καλά προγράμματα, αλλά που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να υποστηριχθούν αν είναι ποιοτικά, προσπαθούμε να πάρουν ένα πιστοποιητικό για να περάσουν στα ευρωπαϊκά ε, και επενδυτικά ταμεία. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε επίσης την εφαρμογή Δηλαδή, ο κόσμος που δουλεύει στις χώρες και στις περιφέρειες να επιταχύνει τις εργασίες, ούτως ώστε να αρχίσουν να λειτουργούν τα προγράμματα, κυρίως να επιλεγούν καταρχήν για να αρχίσουν να λειτουργούν. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα θέματα που ε, θέτονται σε σχέση με τις καθυστερημένες πληρωμές να ρυθμιστούν. Και να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες στις διάφορες περιοχές, βασιζόμενοι στις, ε, στα ΣΥΝ και στις ε, στα πλεονεκτήματα της κάθε περιφέρειας, να υποστηρίξουμε επίσης τις περιοχές και τις περιφέρειες που καθυστερούν. Ειδικά τις επιχειρήσεις που δεν είναι τόσο καλές όσο θα μπορούσε να είναι. Να δούμε τι άλλα εργαλεία έχουμε για να τις βοηθήσουν. Σε σχέση με, τις, με την μακροπεριφερειακή στρατηγική, Επίσης σημειώνουμε το σημείο που, υπόθηκε, που ακούστηκε. Ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια της σημερινής μεταναστευτικής κρίσης. Συνεργαζόμαστε όσο μπορούμε πιο στενά με τις διαχειριστικές αρχές, ούτως ώστε να τις ενθαρρύνουμε να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό, ιδίως μέσα στο τοπικό και περιφερειακό πλαίσιο που τους είναι και πολύ οικείο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νταμάτο έχει το λόγο τώρα για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Θα κάνω και εγώ ίδια τροπολογίες, ούτως ώστε να βελτιώσω ακόμα περισσότερο την έκθεση ε, και περιμένω τις δικές σας. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση που μου έκανε ο κύριος Φανίστελρόι. Ρόι. μια απαρχή απάντηση που μπορώ να σας δώσω για την ερώτηση που μου κάνατε. Το γιατί δηλαδή σε κάποιες χώρες θα πάμε καλύτερα σε σχέση με άλλες στον τομέα των ΜΜΕ ε, στα πλαίσια του θεματικού στόχου 3, η απάντηση θα μπορούσε να είναι η εξή. Γιατί σε ορισμένες περιφέρειες και ορισμένα κράτη-μέλη τα έχουν περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα για τον επιχειρησιακό στόχο 3 που εντάσσονται στον επιχειρησιακό στόχο 3. Μια πρώτη απάντηση και μετά θα δω ε, και τις λεπτομέρειες για να πιστώ ότι όντως αυτή είναι η απάντηση. Επίσης, τις άλλες παραγράφου, τις άλλες ε, παρατηρήσεις για αυτά που είπε ο κύριος Τσίκου εσωτερικοποίηση με καλύτερη, αλλά χω, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της εσωτερικής αγοράς. Αυτό σημαίνει καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών των κρατών μελών, δηλαδή για την ποιότητα των προϊόντων, προϊόντων των επιχειρήσεών μας. Φυσικά, δέχομαι αυτό που είπατε να εντάξω ή μάλλον να αναφέρω καλύτερα το θέμα της ε, κατάρτισης των νέων και να διευκολύνω την ε, γυναική επιχειρηματικότητα που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα σε ορισμένα κρατημέλη. Τι άλλο να πω. Κοινωνική καινοτομία. Ο κύριος Κοντζολίνο το τόνισε αυτό. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις πολύ συχνά σε περιφέρειες με μεγάλες δυσκολίες γίνονται πραγματικά υποκατάστατα του κράτους. Γιατί βοηθούν κατηγορίες ε, ευπαθών πολιτών. Έχουν μεγαλύτερη σημασία λοιπόν στην, ε, στην περιοχή τους, το να δραστηριοποιούνται αυτές οι επιχειρήσεις. Στις επόμενες συνεδριάσεις, λοιπόν, πιστεύω ότι θα κάνουμε μαζί μια καλή δουλειά προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν τη συζήτηση για την εφαρμογή, για την έκθεση εφαρμογής καλύτερα και μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα της ε, πρωίας που είναι το σχέδιο έκθεσης για τις στρατηγικές έρευνας και ανάπτυξης για μια ευφυά εξειδίκευση. Όλα αυτά είναι τμήματα της πολιτικής συνοχής 2014-2020, υποστηρίζουν την θεματική συγκέντρωση και την καλύτερη χρησιμοποίηση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να βελτιώσουν την ε, απόδοση και την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Βασίζονται στις ε, ικανότητες και τα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και ο στόχος είναι να προωθήσουν την ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση όχι μονάχα στις ανεπτυγμένες περιοχές αλλά και σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Όπως αναφέρεται στον κοινό κανονισμό, οι εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές εξειδίκευσης είναι εξάντε αιρεσιμότητα για την χρηματοδότηση από, για τα θέματα αυτά. Τα κάτι μέλη που δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί στο επίπεδο αυτό, συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της Κομισιόν στα θέματα αυτά. Ο κύριος Βαλκαρθέλ είναι ο εισηγητής μας και η προ... προθεσμία για τις τροπολογίες προτείνω να είναι η 5η 25η Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Και έχουμε χρόνο μέχρι τις 10.45 για την συζήτηση αυτή. Κύριε Βαλκαρθέλ, σας δίνω το λόγο <clears throat> και μπορούμε μετά να συνεχίσουμε με τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος γιατί ούτως ή άλλως νομίζω ότι στην ε, παρουσίαση που κάνατε έχετε δείξει περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για ένα θέμα μεγάλης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέμα μεγάλη σημασίας γιατί η καινοτομία αυτή καθεαυτή είναι φυσικά ένα θεμελιώδης θέμα για να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ πιο ανταγωνιστική την οικονομία μας, για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, ποιότητας και να μπορέσουμε να προωθήσουμε με τον τρόπο αυτό την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αλλά επιπλέον, με τα τωρινά λειτουργικά προγράμματα τα οποία είναι σε λειτουργία αλλά δεν έχουν ακόμα συγκεκριμένα αποτελέσματα, η έκθεση αυτή προσπαθεί να φέρει στο φως μερικές βασικές πτυχές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ορισμένες στρατηγικές τόσο για τους δημόσιους φορείς αλλά και για τους ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Επανέρχομαι στο ότι εδώ είναι η πρώτη έκθεση που εκδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας και την έχω διαιρέσει σε έξι τμήματα σαφώς διακεχωρισμένα που για μένα είναι οι κυριότεροι στόχοι <clears throat> δράσης και προώθησης που πρέπει να γίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις στρατηγικές εφιούς εξειδικευσής. Το κείμενο φυσικά θα βελτιωθεί με τις συμβολές και συνεισφορές όλων σας και με απόλυτα πεπισμένος ότι είσαστε όλοι έτοιμοι να βοηθήσετε να εμπλουτίσετε αυτό το κείμενο. Παραμένω λοιπόν να ακούσω τις απόψεις σας στην τωρινή ανταλλαγή απόψεων και με την βεβαιότητα ότι όλοι μας μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα κείμενο το οποίο θα ενισχύσει τις στρατηγικές εφιούς εξειδίκευσης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν για τη βελτίωση αυτού του εγγράφου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Βαλκάρθελ. Ξεκινούμε με τους σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Βανίλτεμπορκ έχει το λόγο. Eh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν ε, άλλοι σκιώδεις ε, από άλλα κόμματα για να παίρνω πρώτο το λόγο. Ε, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή γιατί είναι πολύ ωραία η έκθεσή του, η γνωμοδότηση μάλλον. Έχω κάποιες μερικές λίγες παρατηρήσεις. Προβλέπεται για τα ευρωπαϊκά διορθωτικά ταμεία ένα μεγάλο ρόλο για την καινοτομία. Αλλά στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές δεν έχουμε τέτοια ε, κονδύλια, ούτε είναι μοχλό σε καμία περίπτωση για περισσότερες επενδύσεις στην καινοτομία. Για παράδειγμα, στην Νότια Ολλανδία, από εκεί που προέρχομαι εγώ και κατάγομαι, ε, έχουμε ε, από το Περιφερειακό Ταμείο 75 εκατομμύρια ευρώ μόνο για την προγραμματική περίοδο μέχρι το 2020. Για 7 χρόνια 75 εκατομμυριάκια έχουμε. Αν δείτε ε, τα 3,5 δις που πάνε ετησίως στην έρευνα και την ανάπτυξη, το 90% είναι ιδιωτικές επενδύσεις. Καταλαβαίνετε για ποια τάξη μεγέθους μιλάμε και για ποια προοπτική και υπάρχει μεγάλη σημασία να παραμείνει η ευελιξία δεδομένη ε, για την έρευνα και την ανάπτυξη. Άρα θα πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση ε, συγκεκριμένη ε, με κανόνες και ελέγχους και όχι ένα μοντέλο για όλους. Χρειάζεται διαφοροποίηση. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ περιφερειών. Ε, οι ε, εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με το RIS 3 λένε ότι είναι πάρα πολύ θεωρητικά αυτά τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται και προσεγγίσεις και όταν είναι τόσο θεωρητικά ε, και θέλουμε ευελιξία δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ιστορία 3. Άρα θα πρέπει να γίνουν αλλαγές γιατί αλλάζει η τεχνολογία και αλλάζει και ο κόσμος. Επίσης, θα πρέπει να μειωθούν οι άχρηστες και περιττές διαδικασίες και το γραφειοκρατικό άχθος. Ε, ο καλός ο έλεγχος, καλή η παρακολούθηση, αλλά θα πρέπει να γίνεται με το σωστό τρόπο και θα πρέπει να βελτιώνονται οι φυστάμενοι μηχανισμοί. Με το λεγόμενο Community Innovation Survey που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και είναι μια ε, καλή πρωτοβουλία. Στην παράγραφο 14 ε, γίνεται λόγος για τις διασταυρωμένες ε, επενδύσεις ε, για διασταυρωμένη επικονίαση μεταξύ διαρθωτικών ταμείων και ταμείων στρατηγικών επενδύσεων. Υπάρχουν δυνατότητες με διαφορετικά ταμεία, με διαφορετικά επιτόκια, με διαφορετικό χρόνο κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να μην ε, ασχοληθούμε επιπόλαια με αυτή την προσπάθεια, αλλά σε βάθος και σοβαρά. Ε, η συνέργεια δεν είναι αυτός σκοπός. Η συνέργεια πάντα υποστηρίζει κάποια ε, πολιτική που είναι προσανατολισμένη στην καινοτομία και στην εισαγωγή του στην αγορά. Γιατί πολύ συχνά ο κόσμος πιστεύει ότι από τη στιγμή που θα επενδύσει στην έρευνα και την ανάπτυξη θα βρει ένα καινοτόμο προϊόν. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Χρειάζεται να συνεργαστούν διάφοροι τομείς, χρειάζεται να υπάρχουν ε, στην περιοχή σου κάποιες εταιρείε κλειδιά και κάποιες οικονομικές δομές για να καινοτομείς και να γίνει αυτό προϊόν. Γι' αυτό ε, οι περιφέρειες δεν δεν μπορούν να αντιγράφουν ε, άλλες περιφέρειες για να πετύχουν. Η κάθε μια είναι μοναδική. Αυτό που έχει σημασία είναι να συνεργάζονται και με την ευρωπαϊκή στήριξη να ε, χτίσουμε ερευνητικά κέντρα ως άλλους καθεδρικούς ναούς εν τη ερήμο για να μπορέσει η καινοτομία να βοηθήσει και το οικοσύστημα και τη γνώση να βρούμε τις σωστές εταιρείες να ενισχύσουμε και ε, η γνώση να γίνει προϊόν και το προϊόν να γεμίσει τα ταμεία του ε, καταστήματος. Εκεί χρειάζονται επενδύσεις λοιπόν και στο ανθρώπινο δυναμικό, όχι μόνο στις εταιρείες. Πολλές εταιρείες έχουν πρόβλημα να κρατούν ε, προσωπικό με καλά ε, προσόντα και δεξιότητες. Και άλλες εταιρείες δεν βρίσκουν να προσλάβουν αυτούς που τους χρειάζονται. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν πρόκειται για αυτό το σημαντικό εργαλείο όπως είναι το RIS 3, πρέπει να προωθούμε την καινοτομία που είναι πάντα στην υπηρεσία του ανθρώπου και της κοινωνίας. Ευχαριστώ. του κυρίου Πορέμπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από την πλευρά της ε, συντηρητικής και μεταρρυθμιστικής ομάδος έχουμε μερικά σχόλια. Η ομάδα μας, η ECR, χαιρετίζει την έκθεση αυτή, θεωρεί ότι είναι καλά εδρεωμένη στην κοινή λογική και έχει μια προσέγγιση η οποία είναι επικοδομητική. Συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι πρέπει να υπάρξει έμφαση για στρατηγικές που οδηγούν σε μια ανάπτυξη που βασίζεται σε ευφύη εξειδίκευση και όχι μονάχα σε ανεπτυγμένε περιοχές αλλά και σε περιοχές σε μετάβαση και αγροτικές περιοχές που υπολείπονται σε ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι η ευφύης ε, εξειδίκευση θα πρέπει να είναι μια διαδικασία ανακάλυψης του επιχειρήν με πλήρη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Πρέπει να είναι διαδραστική και να οδηγείται από τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε περιφέρειας και επομένως απαιτεί μια καλύτερη διαδικασία συνεργασίας όλων των επιπέδων κυβέρνησης. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε λοιπόν καλύτερη χρησιμοποίηση των πόρων και ασφάλεια στον τομέα της χρησιμοποίησης ενέργειας και έτσι να αναπτύξει και να απελευθερώσει το αναπτυξιακό δυναμικό κάθε περιοχής και να μπορέσει να φτάσει μια κρίσιμη προσαρμοστική μάζα. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι οι διαδικασίες οι οποίες συνδέονται με αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να απλοποιηθούν και να αφαιρεθούν τα σημεία συμφόρησης για τη στρατηγική αυτή. Κλείνοντας, να σας υπενθυμίσω το ιστορικό αυτής της διαδικασίας. Υπήρξαν ορισμένες ε, ε, σχέσεις μεταξύ βιομηχανιών και των ε, τομέων υποστήριξης σε προηγούμενους αιώνες, αλλά υπήρξαν δυσκολίες στο παρελθόν, γιατί δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα σε ορισμένε περιφέρειες με την αλλαγή της τεχνολογίας ή του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, όπως παραδείγματος χάρη με την εξόριξη άνθρακος ή την αυπηγική. Η ευφύης λοιπόν εξειδίκευση, το να εξειδικεύεται κανείς μόνο σε ένα συγκεκριμένο εγχείρημα και σε ένα τομέα και να συγκεντρώνει εκεί πέρα εξειδικευμένο προσωπικό και εργαζόμενους, αυτό μπορεί να έχει και να επέχει και κινδύνους. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην προσαρμοστικότητα που ανέφερε τώρα ο συναδέλφός μου σε ό,τι αφορά να έχουμε μια εξειδίκευση η οποία είναι εύκαμπτη και προσαρμόσιμη και δεν μας περιορίζει σε σχέση με την ε, χρήση αυτών των δεξιοτήτων. Κατάλληλα όμως πως βλέπουμε σε μια θετική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω και εγώ κάτι για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή εστιάζει βέβαια στην έρευνα και την ανάπτυξη, την ευφυά εξειδίκευση, η οποία όμως περιλαμβάνει ένα ευρύτερο πεδίο του επιστητού και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας να λάβουμε υπόψη μας όλες λοιπόν τις εξειδικεύσεις και τις δεξιότητες που υπάρχουν στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης. Λέμε πάντα ότι οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μοχλή ανάπτυξης. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω το τμήμα της έκτασης που λέει ότι τα διάφορα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές για την ευφυά εξειδίκευση αναγνωρίζοντας τις περιφερειακές πτυχές τους. Μπορούμε έτσι να εξασφαλίσουμε σε καλύτερη χρήση των κονδυλίων συνοχής. Πιστεύω λοιπόν ότι ορθώς η έκθεση αυτή υπογραμμίζει ότι οι στρατηγικές για την εφιούς εξειδίκευσης απαιτούν μια συνέργεια μεταξύ διαφορών κονδυλίων και ταμείων που δεν έχει εξασφαλιστεί μέχρι τώρα. Αυτό απαιτεί, καλύτερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε να βελτιώσουμε αυτή τη μορφή διακυβέρνησης. Πρέπει επίσης να εστιάσουμε και στις μακροπεριφέρειες. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα στην ε, ΕΦΙΑ εξειδίκευση μέσα από μη διαμεθοριακές, μακροπεριφερειακές συνεργασίες ώστε τα σχέδια αυτά να μπορέσουν να εφαρμοστούν καλύτερα και να εξυπηρετήσουν καλύτερα και τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Αυτήν λοιπόν την προσέγγιση θέλω να υποστηρίξω και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή δίνει ιδιαίτερη υπερβολική ίσως ε, Εστίαση στα κέντρα αριστείας. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε όμως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι μοχλή ανάπτυξης. Υπάρχουν και πολλά μικρά πανεπιστήμια στις περιφέρειες της Ευρώπης που μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των περιοχών και με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουν την εφια εξειδίκευση των περιφερειών επί τη βάση των δικών τους ενδογενών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Δεν πρέπει λοιπόν να παραμελήσουμε όλους αυτούς τους πόρους οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν σε επιτυχή προγράμματα. Επίσης ε, δίνει μεγάλη έμφαση η έκθεση αυτή μονάχα στην τεχνική καινοτομία. Ξέρουμε όμως ότι σε πολλά σημαντικά εγχειρήματα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, όπως είναι η κυκλική οικονομία, <clears throat> υπάρχει μια άλλη πτυχή, η επένδυση για τη γνώση των επιχειρηματιών ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν νέα υποδείγματα του επιχειρήν. Είναι σημαντική η κυκλική οικονομία αλλά και η κοινωνική καινοτομία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε μια αλλαγή συμπεριφοράς. Κάτι το οποίο μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα σημαντικό και τα σχέδια που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάποια σχέδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο το έχουν καταδείξει. Δεν μπορούμε να πετύχουμε πολλά αν δεν υπάρξει η αλλαγή της συμπεριφοράς μας και της νοοτροπίας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Πολύ ενδιαφέρον είναι το θέμα. Στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 οι περιφέρειες θα πρέπει να επικεντρώσουν τις επενδύσεις στην έρευνα, κοινοτομία και ανάπτυξη ε, και σε μία έξυπνη εξειδίκευση, λαμβάνοντας υπόψη την εξειδίκευση που έχει κάθε περιοχή. Συμφωνώ ε, με τον συνάδελφο που υπογραμμίζει ότι το RIS 3 θα πρέπει να συνεισφέρει στο να καταστήσει την οικονομία πιο ανταγωνιστική, να δημιουργήσει δηλαδή περισσότερες θέσεις απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εμπειρίες και να διευκολύνει τη διάχυση των, νέων, των βέλτιστων πρακτικών και να ε, μεταλαμπαδεύσει το επιχειρηματικό πνεύμα. Η έμφαση θα πρέπει να δοθεί λοιπόν στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων, των μικρών και των μικρών επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων και στις ε, πράσινε μικρομεσαίες επιχειρήσει και θα πρέπει να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορεί για την εκπόνηση του RIS 3 βασιζόμενοι στην ανάλυση των δυνατών σημείων και στο δυναμικό τη κάθε περιφέρειας. Να επικεντρωθούμε λοιπόν στην, στην παραγωγική εξειδίκευση ούτω ώστε να δούμε τι δυνατότητε έχουμε στα πλαίσια τη έξυπνη εξειδίκευση. Επίση, το RIS 3 με την αρχή της εταιρική σχέσης είναι πολύ σημαντικό το είπε και ο συνάδελφος, ότι στην προετοιμασία αυτή τη περίοδου προγραμματισμού κάποια κράτη-μέλη αποφάσισαν να υιοθετήσουν ε, εθνικά ρίστρια χωρίς να δώσουν στις τοπικές και περιφερειακές αρχές την ε, δυνατότητα να εκπονήσουν τις δικές τους νομοδοτήσεις και επομένως δεν ε, καταλαβαίνουν πραγματικά την σημασία της έξυπνης εξειδίκευσης. και εξάλλου η συνεισφορά των αρχών αυτών θα μπορούσε να βελτιώσει πολύ καλά το πλαίσιο του ΡΙΣΤΡΙΑ. Επίσης, ο συνάδελφος μιλάει για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Γενικά, δεν μπορώ να πω ότι είμαι αντίθετη, αλλά οι τρόποι εφαρμογής θα πρέπει να αξιολογηθούν πολύ ε, προσεκτικά και να παρακολουθηθούν. Αναπερίπτωση ούτω ώστε να μην ε, προωθήσουμε αυτό που έγινε σε, κά, σε κάποιες χώρες, δηλαδή την ε, ιδιωτικοποίηση των κερδών και την, δημο, ε, και την, το να μοιραστούμε όλοι μας τι τις ζημίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έθριτς. Ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή είναι παράδειγμα του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα έπρεπε να το κάνει. Ε, α, περισσότερο σχεδιασμός. Ε, από το 2020 και μετά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα υπερκράτος. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα λεφτά για την έρευνα, αν θέλαμε. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να το κάνουν. Μιλάτε για την ενθάρρυνση της έξυπνης εξειδίκευσης σε ορισμένες περιοχές. Αυτό θα γινόταν με την ελεύθερη αγορά χωρίς να παρεμβαίνετε εσείς. Δεν χρειάζεται κανένα να ξαναγκάσει κάτι. Εγώ εκπροσωπώ το, τα δυτικά Midlands και με ενδιαφέρει ε, το καλό της περιοχής μου και όχι το υπόλοιπο τι, τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Δεν θα μας, δεν θα μας ωφελήσει σε καμία περίπτωση αυτή η προσπάθεια του ΡΙΣ3. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκθεσία όσο και χρήσιμη υπήρξαν πράγματα που θεωρώ και εγώ σημαντικά. Για παράδειγμα, καλύτερο συντονισμός των διαφόρων επιπέδων ε, διαχείρισης, συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μέσων, πηγές χρηματοδότησης, της καινοτομίας κτλ. Θα ήθελα όμως να σας πιστήσω την προσοχή σε ένα σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τις περιφερειακές στρατηγικές για την καινοτομία. Αν το δούμε από αυτή τη σκοπιά, θα διαπιστώσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η ευφυής εξειδίκευση επικαλύπτεται σε διάφορες περιφέρειες με άλλα θέματα. Και είναι πολλές εκείνες οι περιφέρειες που ποντάρουν σε τομείς ε, που είναι του σειρμού, της μόδας και δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις ντόπιε ευκαιρίες, αλλά παρασύρονται. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε και να μας προβληματίσει. Πρέπει επίσης να τονίσουμε κάτι που πολιτικά δεν είναι πάντα πάρα πολύ ελκυστικό, και αυτό είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου. Α πούμε, η λεγόμενη λευκή οικονομία. Είναι μια τεράστια ευκαιρία. Πρόκειται για τη χημική βιομηχανία ή βιομηχανία ε, κατασκευής εργαλειομηχανών, ε, μηχανημάτων. Εκεί δεν υπάρχει πολύ μεγάλη καινοτομία. Ε, και η ευφύης εξειδίκευση αφορά την ανάπτυξη και περιοχών της υπαίθρου και έχει και θέση και χώρο και αξίζει υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνω κι εγώ κάποιες τροπολογίες. Για παράδειγμα, θα πρέπει να τονιστεί και να ενισχυθεί ο συνδυασμός της έρευνας και της ανάπτυξης με τις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής οικονομίας διότι αυτή τη στιγμή κανείς κατανοήσει τον κόσμο της επιστήμης και τον κόσμο της επιχείρησης ταυτόχρονα, αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Υπάρχουν και οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και που διαχειρίζονται τα κονδύλια και θα πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερο θάρρος. Δηλαδή δεν είναι απλοί ταμείες αυτοί, ε, κάνουν και αξιολόγηση, αλλά καλό θα ήταν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να εκτιμούν σωστά τις ανάγκες και να προσπαθούν να καθοδηγούν κάπως ε, τον κόσμο για το ποιες είναι οι δυνατότητες και οι δράσεις που ανοίγονται και οι πιο ελπιδοφόρες δεν μπορούν να έχουν ένα απλό λογιστικό ρόλο ή να μιλούν για μεγάλα έργα και να... Λέιζερ, ξέρω εγώ, ή τέτοια πράγματα, οπτικές ίνες. Αλλά, παρακαλώ, θυμηθείτε ότι πολλές καινοτόμες ε, εφευρέσεις έρχονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στη συνέχεια αναπτύσσονται και γίνονται πολυεθνικοί όμιλοι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανίστελ Ρόε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. έκθεση του συναδέλφου Παλκά Σισό περιγράφει πολύ καλά την κατάσταση. Έχω κάποια σχόλια και εγώ από πλευρά μου. Καταρχάς, αυτό που είπε ο κύριος Έθεριτς, ε, για να βάλουμε τα πράγματα στο όνομα, ε, με το όνομά του για τα δυτικά ε, Midlands είπε ότι από εκεί ξεκίνησε ε, ε, η βιομηχανική επανάσταση. Μιλάτε για την εποχή του λίθου, <laughs> τι ακριβώς αναφέρατε. Η Ευρώπη είναι σε μια τελείως νέα φάση. Δεν μπορεί κανείς να αναπτυχθεί μόνος του, ούτε να αναπτύξει και να εφεύρει νέα προϊόντα και νέα γνώση να μεταφέρει στην πράξη και στην παραγωγική διαδικασία μόνος του. Ταυτόχρονα γίνονται διάφορα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο τον οποίο ζούμε. Και υπάρχει ένας συνδυασμός πληροφορίας και ε, συνεργασίας και στα Midlands που είστε εσείς που είναι πολύτιμο. Όχι ο καθένας μόνος του και ό,τι του φανεί. Αυτό είναι το σημαντικό στην έκθεση. Εκείνος που επιλέγει, ας πούμε, την ευφύ εξειδίκευση, επιλεγει επιλέγει 45 θέματα που υποστηρίζονται από κάτω προς τα πάνω. Στις διάφορες περιφέρειες, στις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που συνεργάζονται μεταξύ τους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θα φέρει την πρόοδο. Δηλαδή ένας είναι ο τροχός, δεν πάει να τον εφεύρει 40 φορές ο καθένας. Το θέμα δεν είναι κάνει ο καθένα 40 αυτοκίνητα, αλλά ε, πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να προχωρήσουμε ε, και να αποδίδει αυτό. Και κάθε περιφέρεια έχει τα πλεονεκτήματα και τα ατού και μπορεί να τα ε, προβάλλει και να τα αξιοποιήσει. Αυτή είναι μια έκκληση δική μου και αξίζει υποστήριξη στην έκθεση. Τώρα επί της ουσίας να πω κάποια πράγματα. Το Δεκέμβριο η Επιτροπή μας επήγε στο κοινό κέντρο ερευνών. Eh, eh, και είδαμε τι έρευνα κάνουν εκεί και πώς πλαισιώνουν ε, την ευφυή εξειδίκευση και την αντίστοιχη πρωτοβουλία σε διάφορα κράτη-μέλη. Και εκεί αναρωτηθήκαμε το ποτήρι τι είναι άραγε, μισοάδιο ή μισογεμάτο. Η απάντηση ήταν ότι ήταν μισογεμάτο μεν, αλλά υπάρχουν πολλά σημεία κριτικής εκεί και κρίσιμα. Αυτή η καινοτομία και η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ε, ευσταθεί. Και υπάρχει αυτή η εξάντε εκ των προτέρων αρεσιμότητα, οι εταιρικέ συμφωνίες και σχέσεις, όλα αυτά είναι καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να έχει και μια διάρκεια αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι που στην παράγραφο 25 ε, καλεί ο εισηγητής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, κάνει μια ενδιάμεση αναθεώρηση, αξιολόγηση και να διαπιστώσει πριν την έβδομη έκθεση συνοχής, πριν κατατεθεί, να δούμε τι πήγε καλά και τι δεν πήγε. Και πού χωλένουν τα πράγματα και πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και προσαρμογές. Εξού και η σημερινή συζήτηση και η ίδια η έκθεση. Και θέλω να ακούσω σήμερα παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς το φαντάζεται όλο αυτό. Ε, κάναμε και μια μήνυ ακρόαση εδώ, σε τούτη εδώ την Επιτροπή και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και τότε ακούστηκε ότι, κοιτάξτε να δείτε, η ευφυής ε, ε, εξειδικευσή θα πρέπει να είναι μια πάγια και διαρκής διαδικασία. Δεν είναι ένα πυροτέχνημα, αφορά την πολιτική συνοχή, στα περιφερειακά ταμεία και τα συνδέει με τους στόχους για το 2020 και μια σειρά άλλα μέσα και εργαλεία που έχουμε. Αυτά είναι αλληλένδετα. Η πολιτική συνοχή δεν είναι κάτι ξεκάφωτο. Πάρε λεφτά εσύ περιφέρεια και κόψε το λαιμό σου. Δεν, ούτε καν πρόκειται για τα χρήματα, αν θέλετε να τα ακούσετε και αυτό. Ε, είναι ότι να έχει όχι ένα τροχό επειδή τον εφήβρες εσύ, αλλά έχει τέσσερι τροχού, ένα αυτοκίνητο το οποίο να κυκλοφορεί στο δρόμο. Αυτή είναι η Ευρώπη. Ας πούμε, τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία της πληροφορία Πριν από 10 χρόνια η Ευρώπη ασχολείται ακόμα με την Νόκια και τα λοιπά και είχαμε εταιρείε παγκόσμιες. Σήμερα που βρισκόμαστε. Για κοιτάξτε ε, πώς έχει η κατάσταση. Χρειάστηκε πια μια παγκόσμια κλίμακα για να έρθει νέα τεχνολογία και να απορροφηθεί και να κυκλοφορεί. Και τώρα αμερικανικές οι εταιρείε που κυριαρχούν. Πια West Midlands. Ποια δυτικά Midlands, οι ευρω... αμερικανικές εταιρείες είναι πολύ πιο πρωτοπόρες, για να καταλάβουμε ποια είναι η κλίμακα και πώς συνεργαζόμαστε. Και καλά χρηματοδοτικά μέσα, νέος τρόπος προσέγγισης, αυτό χρειάζεται να δημιουργηθεί και αυτό είναι η ευφυής εξειδικευσή. Δεν ξέρω αν πρόκειται τώρα για ε, το ε, ε, Internet of Things, για την τρισδιάστατη εκτύπωση, για συγκεκριμένα νέα ε, δεδομένα. Δεν θα πρέπει αυτά να μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις επειδή δεν ασχολούμαστε όλοι μαζί με αυτά. Αυτά είναι τα θέματα ουσίας και σωστά λέει ο συγγητής να ε, συνδυάσουμε την έρευνα, την υλοποίηση, την εφαρμογή, την εφαρμοσμένη έρευνα, το κάνουμε όλοι στα προγράμματά μας τα επιχειρησιακά και Ξέρετε, τα λεφτά δεν ρέουν αυτόματα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτε προς τις επιχειρήσεις και τις περιφέρειες. Αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται με την εκπαίδευση, με την παιδεία ε, στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Ε, capacity building, δηλαδή εκπαιδεύουμε κόσμο, καταρτίζουμε, έχουμε στρατηγική μακροχρόνια. Αυτά είναι τα πράγματα. Και μάλιστα είναι και προαπαιτούμενα όλα αυτά. Και γι' αυτό χαίρομαι που τα λέει όλα αυτά η έκθεση. Και όπως είπα θέλω να ακούσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το θεωρώ σημαντικό. Πώς τα βλέπει όλα αυτά και τι φρονεί για το μέλλον το 16 θα το χρησιμοποιήσει τη χρονιά αυτή για να ε, αξιολογήσει πού βρισκόμαστε και πώς θα προχωρήσουμε στο, ε, στην 7η έκθεση συνοχής. Με μια ανοιχτή συζήτηση που θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Κάτι που μου λείπει τώρα από την έκθεση είναι η ευρωπαϊκή κλίμακα ε, στα ταμεία μας. Έχουμε συνδιαχείριση αποκεντρωμένη και υπάρχουν και ευρωπαϊκά μέσα όπως ορίζον 2020 όπου υπάρχει κεντρική διαχείριση, όπου αποφασίζουν οι Βρυξέλλες ότι αυτό το πρόγραμμα το θέλουμε και το ενισχύουμε και αυτό το έργο όχι. Αυτός δεν είναι ο δικός μας κόσμος, αλλά στην ευφυή εξειδίκευση υπάρχει δυνατότητα όλα αυτά κάπως να κουμπώσουν και όχι μόνο οι πρωτοπόροι, αλλά και οι πρωτοπόροι και εκείνοι που τους ακολουθούν, να μην μείνουν πίσω σε θεματικές ενότητες, σε θεματικές ε, ε, συνεργασίες, να διευκολύνονται αυτά και να τα προωθούμε. Είναι σημαντικό αυτό για την Ευρώπη. Να μην χάσουμε πάλι ούτε το λεωφορείο ούτε το τρένο. Το τρένο του ψηφιακού κόσμου, ας πούμε, σε μερικά σημεία, γιατί μπορεί να το έχουμε χάσει. και να δούμε πώς ξεδιπλώνεται η νέα τεχνολογία και φτάνει στις επιχειρήσεις, στα σχολεία μας κτλ. Ακόμα δεν έχει χαθεί τίποτα εάν το καταλάβουμε και ε, συνεργαστούμε με τέτοιο τρόπο και τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Μια τελευταία παρατήρηση και πάλι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη ρωτήσω τι γίνεται με τις ευφύης πόλεις. Τι είναι αυτό το smart cities και πώς αυτό συνδυάζεται με την ευφύη εξειδίκευση. Ε, το θέμα αυτό των ευφυών πόλεων έχει να κάνει με την κινητικότητα, με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με τις ενέργειες. Είναι, ήταν μια πρωτοβουλία των δημάρχων πριν από μερικά χρόνια. Αλλά ε, η ίδια είναι η μεθοδολογία που κρύβεται από πίσω. Για ποιο λόγο έχουμε τελείως ξεχωριστή προσέγγιση για τις πόλεις, ευφύης πόλεις και για την ευφύ εξειδίκευση σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί είναι κρίμα πιστεύω. Ε, εντάξει υπάρχει αυτό το θέμα του συμφώνου του Άμστερνταμ που αγκαλιάζει τις πόλεις τώρα και ε, τις εντάσσει στην περιφερειακή πολιτική. Θέλω να ακούσω περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα ακόμα τελευταίο. Επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για τα λεφτά, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό. Στο παρελθόν, που δεν είχαμε e, ευφυή εξειδίκευση, Ε, όταν πάσα σε μια εταιρεία το μόνο που έχει μείνει είναι μια κοπέλα στην υποδοχή και η εταιρεία έχει φύγει. Και εσείς μιλάτε για καθεδρικούς να εν τη ερήμο Εδώ θα πρέπει να γίνουν αυτά, όχι να σηκωθούν να φύγουν οι εταιρείε και απλώς να έχουν μια θηρίδα στην οποία να απευθύνεσαι. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί πρέπει να γίνει η εξειδικευσή και να διευκολυνθεί η λειτουργία και η καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν το έχουμε δει ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Όταν πήγαμε στη Σεβίλη, διαπιστώσαμε ότι η ευφυής εξειδίκευση χρησιμοποιείται πάρα πολύ καλά στην προετοιμασία των προγραμμάτων, στην εξέβρεση εταίρων και στη συνεργασία, αλλά αυτό δεν επιταχύνει τα πράγματα. Δηλαδή κάνουν καλά το σχεδιασμό του προγράμματος, αλλά δεν ε, είναι αρκετά καλή στο να βρουν συνεργασίες και το 2016 αυτό θα πρέπει να το προσέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το, το ζητάει ο συγητής και στην παράγραφο 25 είναι σημαντικό για μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βανίσλε. Θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι δεν μπορεί κανείς να μακρηγορεί περισσότερο και από τους εισηγητές αν θέλουμε όλοι να μπορούν να συμμετέχουν σε μια συζήτηση. Συγγνώμη κύριε Φανίσλερο. Λερό. Τελευταία φορά. Ο επόμενος ο μιλτές ο κ. Ρόντνου. Ρόπε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι βραχύτερος του κύριου Φανίσλερο και φυσικά και του εισηγητού. Όταν διάβασα το σχέδιο έκθεσης, είδα τα εξής. Για πρώτη φορά στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να καταρτήσουν στρατηγικές για να ενισχύσουν την έρευνα και την καινοτομία. Παράδοξο λοιπόν μου φαίνεται το ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν στρατηγικές οι οποίες λειτουργούν μονάχα σε εθνικό επίπεδο και όχι σε περιφερειακό επίπεδο. Μα πώς θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν αυτές οι στρατηγικές και εξάλλου πώς τις ενέκρινε η Κομισιόν. Μήπως θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αυστηρότητα όταν εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε την επίτευξη των στόχων αυτών Μήπως η Κομισιόν θα πρέπει να υπενθυμίσει στις χώρες αυτές που υπέβαλαν τέτοιες στρατηγικές ότι πρέπει να συμπεριλάβουν και τις περιφέρειες και να ζητήσουν από τα κατημέλια αυτά να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους. Αλλιώς θα έρθει το 2020 και πάλι θα λέμε φταίνε τα κάτι μελη γιατί δεν έχουμε πετύχει τίποτα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των πολιτικών περιφερειακού χαρακτήρα κτλ. είναι δυνατόν να μην έχουν θέσεις οι περιφέρεια. Αν δούμε την κατάσταση για, την, για τις ανανεώσιμες ενέργειες. 53% των κρατών μελών παίρνουν ενέργεια από άλλες χώρες. Εδώ υπάρχει πραγματικά ένα ευρύ πεδίο για να δράσουμε. Υπάρχουν κράτη-μέλη, υπάρχουν περιφέρειες που παράγουν τα 80% ουσιαστικά των ανανεωσίμων ενεργειών και οι υπόλοιπε μόνο το υπόλοιπο 15% μπορούμε να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ ε, ενεργοί. Και αυτό το βλέπουμε και στη Λιθουανία όταν γίνονται επενδύσεις μόνο για τις επενδύσεις. Όταν υπήρξαν κάποιες επενδύσεις οι οποίες δεν οδήγησαν σε κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν προσεκτική αντιμετώπιση τα θέματα αυτά. Δίνω το λόγο στους εκπρόσωπους της Κομισιόν. Βόλφ και Μάρξ εδώ. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος από τους δύο θα λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο πάντως ως εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ευρωβουλευτές. Είναι πολύ σημαντική έκθεση ίδιο στην παράγραφο 1 που λέει ότι η έξυπνη εξειδίκευση είναι πολύ σημαντική γιατί συνεισφέρει στους στόχους της, του Ευρώπη 2020. Είναι πολύ σημαντικό και η περιφερειακή πολιτική μπορεί να υποστήριξει έτσι την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα συνεργαστούμε με εσά για την έννοια αυτή. Δίδεται μεγάλη έμφαση σε αυτή την έννοια που πρέπει να δημιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω για να είναι δυνατή, να μην επιβληθεί να βασίζεται στο τι θέλουν να κάνουν οι ίδιες οι περιφέρειες. Συνεργαστήκαμε εσά και με άλλους για το, περιφερειακό, για το κανονιστικό πλαίσιο, τόσο ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Και δώσαμε μεγάλη έμφαση στην ε, διαδικασία προγραμματισμού, τόσο ώστε να εξασφαλίσουμε όσο μπορούμε ότι η έξυπνη εξειδίκευση όντως ε, ε, σωματώνεται σωστά στα προγράμματα. Ξέρουμε ότι δεν έχει τελειώσει η προσπάθεια. Θέλουμε να τελειοποιήσουμε τη διαδικασία, αλλά είναι σημαντικό όλο όσο έχει γίνει μέχρι τώρα. Μπορέσαμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλου να το μάθουν, ότι μέσω τη έξυπνη εξειδίκευση να κινητοποιήσουμε ε, υποστήριξη και πραγματογνωμοσύνη από όλε τι υπηρεσίε τη Κομισιόν για να καταστήσουν πραγματικά λειτουργική την έξυπνη εξειδίκευση. Η Γενική Διεύθυνση ε, Έρευνας και Καινοτομίας, ε, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε, συμμετείχαν και το Κοινό Κέντρο Ερευνών επίσης. Οι εταιρικέ σχέσεις στις περιφέρειες προσπαθούμε να λειτουργήσουν καλά. Έχουμε εμπλέξει και ερευνητές σε αυτή τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης και έχουμε εμπλέξει κυρίως τις, α, ε, τους επιχειρηματίες. Και φυσικά τις περιφερειακές αρχές. Και χρησιμοποίησαμε την υποστήριξή σας την περίοδο μετά το 2007, ούτως ώστε η κοινότητα της έρευνας ε, να έρθει σε επαφή με τις ε, επιχειρήσεις, με τις περιφερειακές αρχές και οι, καθυστερη, οι καθυστερημένες περιοχές, χάρη στην υποστήριξή σας, ε, προσπαθούμε να λειτουργήσουν όσο καλύτερα γίνεται, χρησιμοποιώντας τα διάφορα εργαλεία, όπως το εργαλείο για τις μακροπεριφέρειες και άλλα εργαλεία που έχουμε στην περιφερειακή πολιτική, ούτως ώστε οι εταιρικές σχέσεις να λειτουργούν καλά. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται όλα αυτά, ε, μας δείχνει πώς ε, μπορεί να υπάρξει επιτυχία, πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές, πώς μπορούμε να κατανοήσουμε ε, τα όσα κάνουν οι άλλοι και να τα κάνουμε και εμείς. Ε, το βασικό εργαλείο γι' αυτό είναι η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, η πλατφόρμα που υπάρχει για αυτή, που εμείς στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών δουλεύουμε με το Κοινό Κέντρο Ερευνών στη Σεβίλη για να το χρησιμοποιήσουμε. 170 περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη εμπλέκονται εκεί. Ούτως ώστε η προσέγγιση αυτή για την έξυπνη εξειδίκευση να λειτουργήσει. Τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει από τη στρατηγική αυτή έξυπνη ε, εξειδίκευση στις διάφορες περιφέρειες ε, χρησιμοποιούνται ιδίως ε, η υποστήριξη για τις ανανεώσιμες, η ενεργειακή αποδοτικότητα, νανοτεχνολογίες ε, τις αναφέρω για να σας πω ότι δεν μιλάμε μόνο για, τις, ε, για την υψηλή τεχνολογία, αλλά διατροφικό τομέα ε, και διάφορα θέματα που προκύπτουν από την κυκλική οικονομία και τα προωθούμε. Τα θέματα τα οποία θέτεται ε, θέλουμε να εξεταστούν και να συνεισφέρουμε σε αυτά. Ε, την επόμενη εβδομάδα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. Έχουμε με πρωτοβουλία των περιφερειών που ενδιαφέρονται για αυτή την προσέγγιση. Έχουμε μία εκδήλωση όπου διάφοροι εταίροι συνομιλούν, ε, εγκύπτουν επί διαφόρων ε, θεμάτων. 25 και πλέον περιφέρειες ε, ασχολούνται και συνομιλούν. Ε, υπό την αιγίδα της ε, Ολλανδικής Προεδρίας, ούτως ώστε να καταλάβουμε τα πρακτικά στοιχεία, να εμπλακούν οι επιχειρήσεις, να, επίσης η πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων είναι μια άλλη εκδη, έτσι, πρωτοβουλία, ούτως ώστε να ανταλλαγούν γνώσεις, ιδίως στον τομέα της βιοοικονομίας. Και τέλος Απριλίου θα γίνει μια εκδήλωση σχετικά. Ε, σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Βανί Ρόι για την αναθεώρηση φέτος, γίνεται μια σημαντική συζήτηση, θα γίνει μάλλον την, αρχέ αρχές Ιουνίου, ε, διάσκεψη για τις έξυπνες περιφέρειες, είναι το θέμα, και θα δούμε τι έχουμε επιτύχει μέχρι τότε. Θα αξιολογήσουμε δηλαδή και θα από όλη αυτή την προσπάθεια και θα διδαχθούμε και θα χαρτογραφήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι περιφέρειες μπορούν να προωθήσουν τη διαδικασία αυτή Αυτά για φέτος και είναι πολύ σημαντικά. Τώρα κάποια στοιχεία που προέκυψαν στη συζήτηση. Θέλουμε οι προϋποθέσεις να ληφθούν υπόψη και συμφωνούμε με την απόψή σας ότι δεν είναι μία απλή στήρα νομοθετική προσπάθεια, θα πρέπει να δώσει καρπού στην πράξη. Θεωρούμε ότι όλη αυτή η έξυπνη εξειδίκευση δεν αφορά μόνο την τεχνολογία αλλά και τους παραδοσιακούς τομείς, την υψηλή τεχνολογία, αλλά τους παραδοσιακούς τομείς και πρέπει να δούμε τη δύναμη που έχουν οι διάφορες περιφέρειες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εφιστούμε την προσοχή στη δουλειά που κάνατε εσείς για τις καθυστερημένες περιοχές και συχνά για παραδοσιακούς τομείς που τους αμελούμε και που είναι πολύ σημαντικοί. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι λειτουργεί όσο μπορούμε καλύτερα ε, σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία για τις έξυπνες πόλεις. Γιατί οι πόλεις είναι ο χώρος όπου οι καινοτόμες προσεγγίσεις λαμβάνουν χώρα και μπορούμε λοιπόν αυτά τα παραδείγματα να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα αξιοποιήσουμε και να τα απλώσουμε σε όλες τις περιφέρειες. Καλωσορίζω αυτό που λέει η έκθεση επίσης. Για μία έκθεση το 2017, ούτως ώστε να αξιολογήσουμε τη δουλειά που θα έχουμε κάνει, που είναι τόσο σημαντική για την περιφερειακή ανάπτυξη και για την συνεισφορά των περιφερειών στους στόχους Ευρώπη 2020. Θα, γίνουμε, λοιπόν, θα κάνουμε όντως μία αξιολόγηση το 2017. Ευχαριστώ κύριος Βαλκάρθελ. Έχετε το λόγο αν θέλετε να καταλήξετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους παρενέβησαν για το ενδιαφέρον τους και τη σημασία των παρατηρήσεών τους. Ταυτίζομαι με σας. Ταυτίζονται σχεδόν οι απόψεις μας σε όλα όσα αναφέρατε. Σε αυτή την έκθεση, που χάρη στις δικές σας συνεισφορές θα εμπλουτιστεί περαιτέρω, αναφέρεται η ανησυχία για το θέμα της αναγκαίας ευελιξίας, Συχνά είμαστε πολύ θεωρητικοί. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει βραγμού σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να αποφύγουμε υπερβολική γραφειοκρατία δηλαδή στο μέλλον σε αυτή τη διαδικασία. Η καινοτομία απαιτεί ε, την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. και να μην χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μία για τη δημιουργία ε, προϊόντων κλασικών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν το κατάλληλα ε, ενημερωμένο και διαμορφωμένο με τις σωστές δεξιότητες προσωπικό. Στα σημεία που έχει αυτές, αυτή η έκθεση, η αιτιολογική έκθεση, θα συμπεριλάβουμε κάποιες από τις ανησυχίες σας. Ούτως ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή έκθεση. Εκεί που μιλάμε για τη διακυβέρνηση, την πολυεπίπεδη ε, και τις διάφορες, ε, το, το δυναμικό που πρέπει να δημιουργηθεί. Στο σημείο 6 αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη που αποφασίσανε να υιοθετήσουν το εθνικό οριστρία, δεν έδωσαν τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις. Οι τοπικές αρχές φυσικά θα πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και να μην ε, τις αφήσουμε σε υποδέστερο ρόλο σε σχέση με τα κράτη-μέλη, με το εθνικό επίπεδο. Επίσης μιλάμε για, μια, για ένα στενό συντονισμό που θα πρέπει να υπάρχει σε όλη τη φάση εκτέλεσης, εφαρμογής, ανάμεσα στις, ε, στο RIS 3 και στα επιχειρησιακά προγράμματα. Θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία θα πρέπει να έχουμε καινοτόμες ε, πολιτικές, ούτως ώστε να έχουμε μια διαπεριφερειακή συνεργασία και εντός της περιφέρειας και ε, μεταξύ περιφερειών και μεταξύ περιφερειών διαφορετικών κρατών. Ζητάμε επίσης να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες, να μειωθούν ε, τα σημεία συμφόρησης που υπάρχουν στην, ε, στο διοικητικό επίπεδο της, ε, των στρατηγικών. Τα, τα κονδύλια που έχουν σκοπό την ανάπτυξη των περιφερειών και τα άλλα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συντονιστούν καλύτερα. Πιο κάτω στην έκθεση θεωρούμε ότι μόνο λίγες περιφέρειες ασχολούνται με τις ε, ανανεώσιμες ενέργειες, την βιωσιμότητα, την το ψηφιακό θεματολόγιο και είναι κρίμα που μόνο λίγες περιφέρειες ασχολούνται με αυτά. Και θα θέλαμε και άλλες περιφέρειες να ενταχθούν σε αυτή την πορεία και να χρησιμοποιήσουν τα ταμεία ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, μιλάμε για την ανάγκη οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τους δικούς τους μηχανισμούς παρακολούθησης στα πλαίσια μιας συνεχούς αναθεώρησης της ε, στρατηγικής ΡΙΣΤΡΙΑ. Με βάση το, τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και την διασύνδεση ανάμεσα στις προτεραιότητες αυτές και, την, ε, και τις προοπτικές για την ε, μελλοντική ανάπτυξη. Και δύο τελευταία σχόλια. Ένα για την καινοτομία που πολύ συχνά φαίνεται ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται διάφορες μορφές καινοτομία, αλλά που τελικά ε, καινοτομούν μόνο στο λεγόμενο, βασιζόμενες στις λεγόμενες τεχνολογικές γνώσεις. Σε αυτή την έκθεση ε, υπενθυμίζουμε ότι μια καλή στρατηγική δεν μπορεί να δώσει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα εάν δεν δοθούν ε, υπηρεσίες ε, υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις. Ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να λάβω υπόψη τις απόψεις που ακούστηκαν σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά και μείνετε ήσυχοι, θα εντάξω τις απόψεις σας στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε τη συζήτηση για την έκθεση αυτή. Ναι. Και να σας υπενθυμίσω καταληκτική προθεσμία 25 Φεβρουαρίου το μεσημέρι για την κατάθεση τροπολογιών. Επόμενο θέμα τώρα τη σημερινή διάταξή μα είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Σιμ Κάλλα, τον επικεφαλή τη ομάδα υψηλού επίπεδου, για την απλοποίηση τη πολιτική συνοχή. Κάτι που αναφέραμε πάρα πολλέ φορέ στη συζήτησή μα θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον κύριο Κάλλας και να ανταλλάξουμε απόψη μαζί του. Είναι επικεφαλής της νέας ομάδας υψηλού επίπεδου για την παρακολούθηση της ε, καταβολής τους δικαιούχους ποσών <clears throat> από την ε, πολιτική συλλογή. Γεια σας κύριε Κάλλας. Ο στόχος λοιπόν αυτής της ομάδας ψηλοπέδου είναι να μειώσουμε το άχθος της ε, ε, γραφειοκρατίας και των διοικητικών λειτουργιών για τους ε, δικαίουχους. Στις 20 Οκτωβρίου πέρσι, τα 12 μέλη της ομάδας ψηλοπιπέδου με επικεφαλή στον κύριο Κάλλας συναντηθήκαν με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκπρόσωποι της Επιτροπής Ρέντσι στις συναντήσεις αυτές και αυτή της 1ης ε, και 2 Δεκεμβρίου η ομάδα αυτή υψηλού επίπεδου τόνισε την ανάγκη να υπάρξει καλύτερη προσβασιμότητα στην ε, χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρήσης, μείωση του κόστους διοίκησης και καλύτερη λειτουργία των χρηματοδοτικών εργαλείων. Η Επιτροπή ΡΕΓΙ έχει υπογραμμίσει την υποστήριξή της για αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου, τονίζοντας ότι η πραγματική απλοποίηση μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερη προσβασιμότητα για πολλούς ε, περισσότερους δικαιούχους της ε, περιφέρειας της Ευρώπης. Γι' αυτό χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κύριος Κάλλας να λάβει το λόγο στην Επιτροπή μας και να μας παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματα της εργασίας της ομάδος υψηλού επίπεδου. Έχουμε μία ώρα για τη συζήτησή μας με τον κύριο Κάλλας και θα δώσω καταρχήν το λόγο στον κύριο Κάλλας να παρουσιάσει το έργο της ομάδας υψηλού επίπεδου και μετά θα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις και σχόλια από τα μέλη της Επιτροπής μας ξεκινώντας πάντα με τους συντελεστές. Κύριε Κάλλας, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Με χαρά δέχομαι την πρόσκληση και έρχομαι ενώπιόν σας να σας παρουσιάσω την προκατακτική ε, έκθεση ε, της ε, ομάδας μας υψηλού επίπεδου και σε ευχαριστώ που με καλέσατε. Κυρίες και κύριοι, από το 2004 στο 2010 διετέλεσα αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα απαλλαγής προϋπολογισμού και άλλα τέτοια τεινά. Και, και τότε συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά και σκληρά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Για να μειωθεί το επίπεδο των σφαλμάτων στη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων. Και βέβαια η κακοδιαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων ε, ήταν και παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα για την ίδια τη φήμη και το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση αυτή δεν έχει αλλάξει. Υπάρχουν ακόμα σφάλματα και παραδείγματα κακής διαχείρισης και κακής χρήσης ε, των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων που δεν πιάνουν τόπο. Ε, απειλούν το κύρος και τη φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μένα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για να πληστεύσουμε τους κανόνες, να έχουμε λιγότερους κανόνες, λιγότερες επιπλοκές και περιπλοκές, πράγμα που σημαίνει τελικά λιγότερα σφάλματα και περισσότερη διαφάνεια. Βέβαια, αυτό είναι εύκολο να το λες, αλλά πολύ δύσκολο να το κάνεις. Ε, πολλοί δικαιούχοι Μάλλον να το πω αλλιώ. Ποια είναι η εντολή μας. Να ακούμε κυρίως τους δικαιούχου ω ομάδα ε, υψηλού επίπεδου και κάπως να ακούμε ε, τη γνώμη τους και να τις ε, συνδυάσουμε και να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Και διαχειριστικές αρχές και οργανισμοί, όλα αυτά θα πρέπει να δίδονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω ε, διαβουλεύσεις και παρατηρήσεις. Πολλοί δικαιούχοι ε, παραπονιούνται ότι είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ακόμα και όταν φτάσουν μετά η διαχείριση των έργων με όλη τη γραφειοκρατία και τα συμπαρομαρτούντα και τα παρελκόμενα ε, τους κάνουν τη ζωή δύσκολη. Βεβαίως αυτό είναι κακό και θα πρέπει να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να το διορθώσουμε. Βασικός μας στόχος λοιπόν είναι να εξασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε όλα τα εδεχόμενα και τις δυνατότητες να πλουστεύουμε τη ζωή των δικαιούχων. Και τα κρατημέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνουν αυτό. Κοιτάξαμε και θετικά παραδείγματα για το πώς γίνεται ήδη κάτι τέτοιο και τους λόγους για τους οποίους ε, άλλοι διστάζουν να το κάνουν. Ε, θα πρέπει να βρούμε λοιπόν νέους τρόπους απλούστευσης. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα τις πρόσφατες συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απλοποίηση και προτίθεμαι να συνεισφέρει η ομάδα μας με τρόπο ενεργό στη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ζήτησε να κάνουμε συστάσεις για συγκεκριμένες δράσεις και μετά να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό απλοποίησης ε, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Από τώρα δηλαδή. Ε, σε αυτό εστιάζουμε, που είναι η περίοδος 2014-2020. Βεβαίως κοιτάμε και το διάστημα μετά και επέκεινα. Αλλά θα έρθω σε αυτό λίγο αργότερα. Ε, τα αρχικά λοιπόν συμπεράσματα ποια είναι και οι συστάσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου. Ήδη αρχίσαμε να μελετούμε σε λεπτομέρειες τέσσερα θέματα το Δεκέμβριο. Ε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, απλούστευση κόστος, ε, πρόσβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κοινοτική χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά μέσα. Έχουμε εισηγητές που εργάζονται για τα συμπεράσματα και τις συστάσεις και στις αρχές του μήνα, ε, εκτός από το Δεκέμβριο, συζητήσαμε και θα δημοσιευθούν όλα αυτά μέχρι τέλη Φεβρουαρίου και τα υπόλοιπα ε, μέχρι το καλοκαίρι. Σήμερα θέλω να σας δώσω μια μυρωδιά από τις βασικές συστάσεις και τα συμπεράσματα που συζητούμε. Ε, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη την επόμενη περίοδο να έχουν μια κοινή πλατφόρμα ή σύστημα για τη χρηματοδότηση, ε, για τους δικαιούχους, για τον έλεγχο και την πληροφορία και τη τεχνολογία της πληροφορίας. Για τη σημερινή προγραμματική περίοδο χρειάζεται να γίνει προσπάθεια για να μην υπονομευθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και να απλουστευτεί η διαχείριση των ταμείων και να απλουστευτούν οι διαδικασίες για να μπορούν να ζητούν χρηματοδότηση και την αντιλαμβάνουν οι δικαιούχοι. Αυτό πώς θα γίνει. Να γίνονται καλύτερα δεκτά τα ηλεκτρονικά έγγραφα για όλα τα ταμεία και ε, ε, χρειάζεται καλύτερο έλεγχο και μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο να ενέχεται. Τι μπορώ να σας πω για τη συζήτηση αυτή. Έχω ακούσει ε, πάρα πολλές εμπειρίες και προηγμένες σε πολλά κρατημέλη και μεταξύ ε, Αυτή είναι η πατρίδα μου που ε, είναι περήφανη για την ηλεκτρονική της διακυβέρνηση. Αυτό δεν είναι θαύμα, γίνεται. Υπάρχουν όμως ζητήματα για τη λήψη των αποφάσεων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρέπει να λυθούν, που πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστούν. Έτσι. Η ηλεκτρονική διαχείριση λοιπόν και διακυβέρνηση είναι κάποιος πιο περίπλοκη γιατί είναι πιο ευάλωτη σε κάποιες αλλαγές που γίνονται. Ιδιαίτερα όταν αλλάζεις τους κανόνες χρειάζεται μια συγκεκριμένη ανάπτυξη που θέλει και το χρόνο της για να αναπτυχθούν λύσεις ε, πληροφορικής. Και υπάρχει και ένα ζήτημα συμβατότητας διαφόρων λύσεων ε, πληροφορικής, ε, η ακαιρεότητα των δεδομένων, η αποθήκευσή τους, η εξασφάλισή τους και το μεγάλο θέμα της ασφάλειας ε, της πληροφορικής, το οποίο το συζητούν πολύ και σε πολλά επίπεδα. Και υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Υπάρχει ένας αναλφαβητισμός από πλευράς δικαιούχων ως προς την πληροφορική και θέλουν και ειδική κατάρτιση οι ίδιοι για να διαχειρίζονται τα προγράμματα αυτά και τα έργα, πράγμα που σημαίνει επιπλέον προσπάθεια, κόπο και κόστος ε, σε σχέση με το πιθανό όφελος. Αλλά όταν λειτουργούν αυτά τα εργαλεία της πληροφορικής ε, είναι πολύ πιο εύκολο και υπάρχουν πολλά ωφέλη και για τους δικαιούχους τους ίδιους και πρέπει να το καταλάβουν. Όταν έχει ε, κάποιος τη δυνατότητα να το κάνει είναι καλύτερο. Λοιπόν, το κόστος να είναι πιο ε, απλό ή μάλλον οι δυνατότητες να είναι απλουστευμένες, ιδιαίτερα όταν έχουμε σύγκρουση με άλλους κανόνες όπως είναι οι κρατικές ενισχύσεις. Ε, θα πρέπει το συντομότερο αυτά τα θέματα να λύνονται και δια της νομοθετικής οδού και με νομοθετικές προσαρμογές. Οι απλουστευμένες λοιπόν ε, επιλογές κόστους βασίζονται πάντα σε αποτελέσματα και όταν φτάνουμε στα αποτελέσματα αυτά ε, χρειάζεται υποστήριξη εκ των προτέρων ε, για τις δομές αυτές για να ξέρουμε τι δυνατότητες υπάρχουν από την αρχή. Ε, όπως αναφέρονται και στον αντίστοιχο κανονισμό. Και θα πρέπει πιο γρήγορα να εγκρίνονται οι διάφορες μέθοδοι που αναπτύσσουν οι αρχές που διαχειρίζονται τα έργα. Η πρόσβαση στην κοινωτική χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες. Έγινε μία πρώτη μόνο συζήτηση, αλλά φαίνεται ότι και εδώ χρειάζεται απλούστευση, να μπορούν πιο εύκολα να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια και να είναι και πιο ελκυστικά αυτά όλα για τις μικρομεσαίες. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται πιο συνεκτική προσέγγιση και να είναι στο κέντρο της διαδικασίας οι πραγματικές ανάγκες. Αυτό φαίνεται να λειτουργεί όταν τα κράτη-μέλη είναι προσιλωμένα σε αυτή την ε, προσπάθεια και έχουν στόχους για τη μείωση του διοικητικού άχθους. Και επίσης από τις πρώτες συζητήσεις το πρόβλημα που έχουμε για τα χρηματοδοτικά μέσα φαίνεται να απορρέουν ότι, από το γεγονός ότι οι δικαιούχοι έχουν ένα γολγοθά να ακολουθήσουν και διοικητικό και πληροφοριών αντίστοιχο με εκείνο των επιδοτήσεων. Ε, δηλαδή ε, είναι πολύ βαριά η διαδικασία. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάγκη για μια πιο ευέλικτη προσέγγιση για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά εργαλεία χρηματοδοτικά διαφορετικής φύσεως. Εδώ θα χρειαστούμε περισσότερες συζητήσεις για να αντιμετωπίσουμε την πολυπλοκότητα των θεμάτων αυτών και τώρα θα ήθελα να σας κάνω μερικά σχόλια περαιτέρω που θα μπορούσαν να είναι έναρσμα για περαιτέρω αναστοχασμό και προβληματισμό μεταξύ των λιπτών απόφασης στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο. Έχει αυξηθεί βέβαια η πολυπλοκότητα των κανονισμών. Είναι ακόμα πιο μακροσκελής κανονισμοί από ό,τι στο παρελθόν. αυτή τη στιγμή έχετε πέντε ευρωπαϊκές δομές ταμείων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων και κάπου 500 προγράμματα τα οποία διαγωνίζονται για την χρηματοδότηση. Και αυτό είναι και πρωτοβουλία των κρατών μελών να δημιουργούν περισσότερα προγράμματα. Αν έχει κανείς περισσότερα προγράμματα πρέπει να είναι και πιο πολύπλοκοι οι, κατα... οι κανονισμοί, κάποιος πρέπει να τους ελέγξει, κάποιος πρέπει να κάνει επιλογή των προγραμμάτων. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ξέρουν όλοι είναι ότι υπάρχει μεν ο κανονισμός που οι κανονισμοί που έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο, αλλά υπάρχουν παράλληλα κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες είναι πολλές, μακροσκελείς και αυξάνονται. 880 κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική συνοχής, για το ταμεία συνοχής. Οι δικαιούχοι λοιπόν <clears throat> λογικά έχουν πολλές αντιρρήσεις για όλες αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Έχουμε να κάνουμε μια διαδικασία που δεν είναι διαχειρίσιμη Όπως είπε κάποιος, είναι μια ζούγκλα κανονιστικών ρυθμίσεων που δεν μπορεί κανείς να βρει την άκρη, είναι ένας κικαιώνας αδιαπέραστος. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλα αυτά και μόνο όταν η Κομισιόν έχει φτάσει σε κάτι ε, θα είναι πιο διαχειρισμή κατάσταση. Αλλά η εμπειρία δείχνει ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές γίνονται ήπια νομοθεσία και τελικά κάνουν ακόμα πιο πολύπλοκη και αβέβαια τη διαχείριση των κανόνων και δημιουργούν και έλλειψη νομικής ασφάλειας. Πολύ συχνά μεταρρυθμίζονται αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές. Σας λέω λοιπόν τι μου μεταφέρουν οι δικαιούχοι στην ε, συζήτηση αυτή που έγινε και τη διαβούλευση. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές, τι νομική βάση έχουν. Είναι ένα είδος παράλληλης νομοθεσίας <clears throat> η οποία δεν έχει περάσει από καμία διαδικασία και ήδη τροποποιούν την νομοθεσία που είναι ήδη πολύπλοκη και μακροσκελής. Και οι δικαιούχοι θα θέλανε να υπάρξει μια καλύτερη λύση για όλα αυτά τα προβλήματα. Ένα σύστημα λοιπόν το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να δίνει λαβές σε αυθαίρετες ερμηνείες. Πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ο λογιστικός έλεγχος. Και έχουν πει όλοι οι δικαιούχοι ότι είναι πάρα πολλά τα επίπεδα ελέγχου που είναι και δυσανάλογα προς τα ποσά τα οποία εμπλέκονται και έχουμε προτείνει να μειωθεί η ανάγκη για λογιστικούς ελέγχους και γενικότερα ελέγχους. Η αβεβαιότητα λοιπόν για τους ελέγχους είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα στους δικαιούχους. Και επίσης αυτό αφορά φυσικά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, αλλά είναι σημαντικά θέματα. Συζητήσαμε λοιπόν με τους δικαιούχους πώς να βελτιώσουμε την κατάσταση, μας είπαν ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκες κατευθυντήρες γραμμές. Υπάρχει αβεβαιότητα σε σχέση με τους λογιστικούς ελέγχους και υπήρξαν και άλλες συγκεκριμένε και ενδιαφέρουσες προτάσεις για την ε, αύξηση του κατοφλίου του ε, ανεκτού ορίου. Ξέρετε ότι αυτό είχε καθοριστεί στα 2%. Αλλά βέβαια από πολιτική άποψη όλα αυτά τα σφάλματα είναι αποδεκτά. Δεν είναι αποδεκτά μάλλον. Η πρόταση λοιπόν να ανεβάσουμε στα 5% το επίπεδο, το κατόφλιο του αποδεκτού σφάλματος είναι δύσκολο να γίνει πραγματικότητα. Πρέπει να γίνουν λοιπόν όλα αυτά για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να έχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα σε σχέση με τα θέματα αυτά. Όλα αυτά είναι απλώς τα πρώτα μας πορίσματα στην ε, διαδικασία της ομάδας εργασίας και όταν είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις, λεπτομεριακές, θα υπάρξει ένα έγγραφο το οποίο θα είναι στη διάθεση όλων. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή και τώρα οι συναδελφοί έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το λόγο. Ξεκινώ με τους συντονιστές, τον κύριο Φανίς ε. ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάρας, με μεγάλη χαρά σας βλέπουμε εδώ ενώπιόν μας. Ξέρω ότι κάνατε μεγάλα βήματα. Θυμάμαι τη συζήτησή μας για την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για τη Διασύνδεση, όπου είδαμε από το Ταμείο Συνοχής την προοπτική και τα ειδικά προβλήματα που είχατε αντιμετωπίσει τότε και κάνατε πολύ μεγάλη πρόοδο. Προς την ίδια κατεύθυνση λοιπόν είναι και η ερώτησή μου για την εντολή σας πρώτα απ' όλα. Ε, σας επιτρέπουν να κάνετε συγκεκριμένες προτάσεις για να αλλάξουν οι κανονισμοί και εσείς το πράτετε ή θα το κάνετε. Γιατί σε πολύ σύντομο χρόνο αναφέρετε πάρα πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς μπορούν να αλλάξουν και ότι πρέπει να αλλάξουν. Δεύτερον, Διαβάσατε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά. And, and Πώς σας φάνηκε. Ε, πήγατε στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να προχωρήσουμε. Στην έκθεση Thomas Deutsch, στην έκθεση για τη συνοχή, είπαμε ότι ως κοινοβούλιο είμαστε πρόθυμοι και προετοιμασμένοι να γίνουν τεχνικές προσαρμογές ε, της ε, τρέχουσας διαδικασίας και του συγκεκριμένου κανονισμού. Συγκεκριμένα για αυτό το στόχο. Όχι να χτίσουμε νέο καθεδρικό ναό πάλι με ρυθμίσεις και κανονισμούς, αλλά να κάνουμε συγκεκριμένες προσαρμογές για να γίνει συγκεκριμένη πρόοδος. Και άκουσα από τον τύπο ότι και στην Επιτροπή ε, Περιφερειών δεν θέλουν αλλαγές τώρα. Ε, το 2018 κύριε Κάλλας ή κάποια στιγμή θέλουν αλλαγές τώρα. Μπορείτε λοιπόν να μας ενημερώσετε τι γίνεται, ε, πώς προτίθεστε να προχωρήσετε και με ποιο τρόπο εμείς μπορούμε να σας ε, βοηθήσουμε. Να πέσει αυτό το όριμο φρούτο για να βοηθήσει τους δικαιούχους επιτέλους. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Το ξέρω ότι δεν θα γίνει κανένα big bang, αλλά να κάνουμε μικρά βήματα ε, τα την παρούσα τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Αυτά. Σοσιαλιστές, ο κύριος Βον. Ευχαριστώ τον κύριο Κάλλας για την παρουσίασή του. Εμείς στην ομάδα μας, μαζί με άλλους ε, συναδέλφους στην με Επιτροπή Ρέτζι θεωρούμε ότι η Επιτροπή που προεδρεύεται είναι πολύ σημαντικό για, την, για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και της περιφερειακής πολιτικής. Συχνά υπάρχουν δικαιούχοι και διαχειριστικές αρχές που μας λένε το ίδιο. Ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος ό,τι αφορά την απλούστευση, αλλά πιστεύουν ότι πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν και είναι κρίμα που δεν έχετε ευρωβουλευτέ στην Επιτροπή σας. Έχουμε και την εμπειρία και τη γνώση για να συνεισφέρουμε στη συζήτησή σας. Ε, θα έπρεπε να βρείτε κάποιο τρόπο για να εμπλέξετε τους ε, ευρωβουλευτέ στη συζήτηση. Σε ό,τι αφορά τις αρχικές συστάσεις που μας παρουσιάσατε, αναφέρατε μία που είναι πολύ σημαντική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για όλους τους δικαιούχους και τις διαχειριστικές αρχές. Να υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση στους ελέγχου. Τις, τις περασμένες εβδομάδες μιλήσαμε για τις ευκαιρίες ε, που θα είχε το να υπάρχει ένας έλεγχος. Το ελεγκτικό συνέδριο βέβαια ε, μπορεί να έχει αντιρρήσει στο να υπάρχει ένας και μόνο έλεγχος. Και οποιασδήποτε προτάσεις για αλλαγή του ελεγκτικού συστήματος, ε, υπάρχουν τους χάρη τους κανόνες προμηθειών, που είναι άλλη προβληματική περιοχή, όλα αυτά τα στοιχεία θα χρειαστεί να συζητηθούν ε, με το ελεγκτικό συνέδριο. Το πρώτο μου ερώτημα είναι, Προβλέπετε τέτοια συζήτηση με το Ελεκτικό Συνέδριο, γιατί κάποια από τα πράγματα που μπορεί να συστήσετε ε, πρέπει να περάσουν και από το Ελεκτικό Συνέδριο. Πρέπει να εγκριθούν από το Ελεκτικό Συνέδριο και αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο που είναι σημαντικό για μα είναι οι κανόνε ε, κρατικών ενισχύσεων. Αναφέρατε τι ε, ευκαιρίε για απλούστευση των κανόνων αυτών. Τι είδου αλλαγέ φαντάζεστε ότι θα λάβουν χώρα. Είναι δύσκολο να το φανταστούμε. Ορισμένοι λένε θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Βεβαίως, αν έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία, αυτό έρχεται σε αντίφαση με το να έχουμε κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Πρέπει να βρούμε κάποια ισορροπία ανάμεσα στα δύο, ευελιξία και κανόνες. Ε, βέβαια, μπορεί να είναι αρχική φάση, αλλά μπορείτε να μας δώσετε κάποιε ε, ιδέες για του κανόνες κρατικών ενισχύσεων που μπορεί να είναι χρήσιμε για μας. Ευχαριστώ, κύριο Λούερ. Μ' αρέσει το σχόλιο που κάνατε για την διαλειτουργικότητα των συστημάτων μηχανοργάνωσης και πληροφορικής. Το ήταν αίτημα των stakeholders και μας ενδιαφέρει πολύ. Επίσης, μεγαλύτερη εστίαση ε, σε μια διαδικασία επιλογής πιο έτσι, επιχειρηματικού χαρακτήρα. Επίσης, ε, για την ήπια νομοθεσία και ποιες είναι οι ανεπιθύμητες συνέπειες αυτής. Ε, πιθανή σύγκρουση επιθυμιών. Από τη μία ευελιξία, από την άλλη όμως θέλουμε και τυποποίηση. Και παράλληλα και απλούστευση. Και παρότι αυτά δεν είναι απόλυτα αντιφατικά μεταξύ τους, υπάρχει ένα δυναμικό να συγκρουστούν. Πώς μπορούμε, να, πώς μπορούμε να τα πετύχουμε και τα τρία χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να μην πετύχουμε τίποτα ε, λόγω του ότι έρχονται σε αντίφαση ή σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ποιες είναι οι ιδέες σας. Επίσης ε, θα θέλαμε η πολιτική συνοχή να ενταχθεί στην πολιτική, στην πρωτοβουλία μάλλον του εφνομοθετή, της καλύτερης νομοθεσίας. Κάποιες ιδέες γι' αυτό. Και τέλος το άλλο που μας ενδιαφέρει είναι πού μπορείτε στα πλαίσια της εντολής σας να δουλέψετε και να βελτιώσετε το πρόβλημα του θέματος της απορρόφησης. Ε, υπάρχουν προβλήματα με την Ελλάδα, ανέκυψαν πρόσφατα, με την Κροατία και με άλλες χώρες, που συνδέεται με την απλούστευση. Εάν δεν έχεις πρόσβαση στα ταμεία, λόγω του ότι έχεις κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, αυτό δημιουργεί δυσκολίες και αυτό, εν συνεχεία, είναι εις βάρος της ε, φήμης ή της ε, ικανότητας των ταμείων να πετύχουν τους στόχους τους. Ε, διερωτώ με αν το αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα, αν το συζητάτε. Αυτή η καθοδήγηση όμως ε, και η τάση προς την ήπια νομοθεσία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η ευελιξία από τη μία ε, σε αντιπαράθεση με την ε, απλούστευση και την τυποποίηση. Πώς μπορούμε να τα πετύχουμε και τα τρία χωρίς να έρθουν σε σύγκρουση και να μην πετύχουμε τίποτα τελικά. Ευχαριστώ κύριος Βαμίλτεμπρουκ από τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς όρισατε κύριε Κάλλας. Και ίσως είναι υπερβολικό να πει κανείς ότι ο κόσμος όλος έχει στραμμένα τα μάτια του σε εσάς και το έργο σας. Πάντως έχει σημασία αυτό που κάνετε και τουλάχιστον ένα κομμάτι της Ευρώπης που ε, ασχολείται με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία περιμένει τις δικές σας συστάσεις γιατί η απλούστευση της πολιτικής συνοχής είναι κομβική για να πετύχουμε την επόμενη περίοδο την πολιτική μας συνοχής. Τρία πράγματα. Ερωτήσεις βασικά. Πρώτη θα κοιτάξετε και τις διαφορές όταν για παράδειγμα συζητούμε για την επέμβαση και παρέμβαση των Ευρωπαϊκών Ταμείων στην ε, περιφερειακή πολιτική, τις διαφορές λέω ε, στη ε, διάδραση του Ιντερεκ με τα ΕΣΠΑ γιατί πολλοί δικαιούχοι διαμαρτύρονται ότι το Ιντερεκ είναι πάρα πολύ ειδικό όταν μιλάμε για το γραφειοκρατικό άχθος γιατί ε, παρεμβαίνουν και διάφορες ε, διοικητικές ε, κουλτούρες και παραδόσεις των διαφόρων κρατών εκεί. Δεύτερη ερώτηση ή σχόλιο έχει να κάνει και πάλι με το γραφειοκρατικό και το διοικητικό άχθος όταν μιλούμε για το λογιστικό έλεγχο. Και αυτό είναι ένα σχόλιο και προς τον συνάδελφό μου. Όταν μιλάμε για το ελεκτικό συνέδριο, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ πρόθυμοι πάντα να έχουν ένα ενιαίο σύστημα λογιστικού ελέγχου που να ισχύει παντού πώς θα αποφύγουμε τη σώρευση ελέγχων και την επικάλυψη και να έχουμε υπερβολικούς ελέγχους και να έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν βασίζεται στην εμπιστοσύνη αλλά στην καχυποψία και στη δυσπιστία. Και ε, το τρίτο και τελευταίο, η απλούστευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλέ φορέ ακούω ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερου κανόνε και σε περισσότερο διοικητικό άκθο σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και εθνικό. Διότι έρχονται να καλύψουν το διοικητικό κενό οι κρατικές διοικήσεις και οι περιφερειακές. Και ο κόσμος δείχνει μια προθυμία να μειώσουν αυτό το γραφειοκρατικό άχθος. Μα πρέπει το σύστημα να βασίζεται στην εμπιστοσύνη, όχι στη δυσπιστία. Από τη χώρα μου βλέπω ότι η μείωση των διοικητικών κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο οδήγησε σε τεράστια αύξηση των εθνικών κανόνων από την Ολλανδία. Πώς το βλέπετε εσείς. Παρακαλώ. Κύριο Σομάζου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κάλλας, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και την παρουσίασή σας. Έχετε μια σημαντική ευθύνη η οποία δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής αλλά συγχρόνως είναι και πολύ πολιτικού χαρακτήρα γιατί ξέρετε σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης οι δικαιούχοι μας λένε «Μα πώς μπορείτε να έχετε φτιάξει ένα τέτοιο πολύπλοκο σύστημα όπως αυτό που έχετε. Γιατί δεν μπορείτε να απλοποιήσετε τους κανόνες. Και είναι πραγματικά πολύ σωστό αυτό. Για την ε, περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 είπατε ότι έχετε περίπου χίλιες σελίδες κανονισμού 7 ειδικούς κανονισμούς, 6 κατεξουσιοδότηση πράξεις, 8 εκτελεστικές πράξεις και 800 κατευθυντήριες. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να καταλάβει κανείς και να, έχει να βρει τον μπούσουλα. Και όλα αυτά βέβαια έχουν και πολύ πολιτικό χαρακτήρα. Γιατί η δυσφορία η οποία δημιουργείται και η απόσταση μεταξύ των λαών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται ακριβώς σε αυτή την αδυναμία κατανόησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της αδυναμίας να μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί στις αιτήσει <clears throat> που στα αιτήματα των ευρωπαϊκών κανονισμών για τα προγράμματα αυτά. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε στην ουσία του θέματος. Και ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω. Πρέπει να αναρωτηθούμε πώς αυτή η Ευρώπη η οποία θέλει να έχει φιλελεύθερες πολιτικές έχει καταφέρει να γίνει αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας που απλώς ενδιαφέρεται για νομοθεσία και περαιτέρω νομοθεσία. Και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε και στην απάντηση αυτού του προβλήματος νομίζω ότι θα βρείτε και την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δικαιούχων πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνη την καχυποψία που οδηγεί πάντα σε διαδικασίες ελέγχου που είναι όλο και πιο άκαμπτες και επαχθείς. Προχθές ήμουν σε μια συνεδρίαση στο Παρίσι για το πρόγραμμα Στρατηγικών επενδύσεων που έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει και να ανταποκριθεί με μεγάλη ταχύτητα στις ανάγκες απασχόλησης και επενδύσεων και οικονομικής μεγέθυνσης. Υπάρχει βέβαια ένα σύνολο στόχων που έχουν επιτευχθεί, αλλά όλοι οι ενδιαφερόμενοι μου είπαν και πάλι ότι να έχουμε και πάλι ένα τεράστιο και πολύπλοκο σύστημα. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα θέματα. Ξέρετε, και το είπατε νομίζω, ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια σε σχέση με τις γλώσσες στις οποίες ε, διατυπώνονται οι κανονισμοί, γιατί υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την μετάφρασή τους και την ερμηνεία τους. Οι κανονισμοί αυτοί και οι ερμηνευτικές διατάξεις να στη διάθεση όλων για να μπορούν να καταλάβουν περί πρόκειται. Και επίσης θα πρέπει να βασίσουμε τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση των μικροτέρων δικαίουχων γιατί οι μεγάλοι δικαίουχοι έχουν τις ικανότητες, τους πόρους τους ανθρώπινους και τους τεχνικούς να αντιμετωπίσουν <clears throat> την πολυπλοκότητα της νομοθεσίας. Αλλά οι πιο μικροί δικαιούχοι, αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν τα μικρά σχέδια, έχουν τεράστιες δυσκολίες με την ερμηνεία των ευρωπαϊκών κανονισμών. Τέλος, όλοι θα πρέπει να υπομισθούν τις ευθύνε τους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης έχει μια μεγάλη ευθύνη ως συνομοθέτης μέσα στα πλαίσια των τριλόγων, όταν συζητούνται τα προγράμματα 2014-2020, εμείς είχαμε τονίσει ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, αλλά στην πράξη έχουμε πολυπλοκοποιήσει ακόμα περισσότερο τους κανόνες. Γι' αυτό το διάστημα 2020-2027 η δική μας ε, ομάδα διαπραγμάτευσης πρέπει να αγωνιστεί για την απλοποίηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν βλέπω τον κύριο Σκλέσσερς. Α, η κυρία Ταμάτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάλλας που ήρθατε. Σας περιμέναμε εδώ και καιρό. Και στην έκθεση του Κοινοβουλίου αυτό διαφαίνεται. Συμφωνώ με το αίτημα άλλων συναδέλφων που αφορά την εντολή που έχει η ομάδα υψηλού επίπεδου σας. Τι σκοπεύετε δηλαδή να κάνετε τελικά. Το 2017, αν κατάλαβα καλά, θα έχετε το καθήκον να ασχοληθείτε με την περίοδο μετά το 2020. Πώς θα το κάνετε, μέχρι ποιου σημείου θα φτάσει η αλλαγή των ε, σχετικών κανόνων μας είπατε ότι εμπλέκονται στην όλη διαδικασία και οι δικαιούχοι. Νομίζω ότι καλό είναι αυτό, η προσέγγιση σας όμως νομίζω ότι είναι από πάνω προς τα κάτω, όχι από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, ποια κατηγορία δικαιούχων ακούτε και με ποια κατηγορία συνομιλείτε. Θα ήθελα να ακούτε μια... Φοβάμαι ότι ακούτε μόνο θέλω μάλλον να ακούτε κατηγορίες ανθρώπων έτσι πιο πολυπληθών ε, και όχι πιο μικρές κατηγορίες. Επίσης, για το e-governance. Πριν το καλοκαίρι, ή μάλλον θα έχετε έτοιμα τα απορίσματα το Φεβρουάριο ε, και για τα τρία άλλα θέματα πριν το καλοκαίρι θα είστε έτοιμοι και θα, έρθετε εδώ πέρα για να λογοδοτήσετε και στην Επιτροπή μας αλλά και στο Κοινοβούλιο. Για τη συζήτηση που αφορά την απλούστευση ε, κάνετε, λαμβάνετε υπόψη σας την ε, εξισορρόπηση του ελέγχου από τη μία και την καταπολέμηση της απάτης από την άλλη. Ευχαριστώ. Αυτέ ήταν οι ερωτήσει των συντονιστών των πολιτικών ομάδων. Θα απαντήσει πρώτα ο κύριο Κάλλε και συνεχεία οι υπόλοιποι ευρωβουλευτέ θα θέσουν τι ερωτήσει του. Ευχαριστώ. Πολύ οικία μου ακούστηκαν κάποια από αυτά τα ερωτήματα. Τα έχουμε συζητήσει στι συνεδριάσεις τη Επιτροπής Ελέγχου των Προπολογισμών. Η σχέση μεταξύ ελέγχου, Φερρυπίν, και αποφάσεων. Είμαστε στην αρχή της ε, προσπάθειάς μας, ε, στην αρχή των εργασιών μας. Ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι τώρα για να ετοιμάσουμε τα συμπεράσματά μας για το e-governance, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και απλουστευμένες διαδικασίες, επιλογές ε, Αρχικά η εντολή μας ήταν διατυπωμένη έτσι ούτως ώστε να παρακολουθούμε το πώς βλέπουν οι δικαιούχοι τη χρήση των ταμείων και την ύπαρξη των κανόνων για τα ταμεία. Δεν πρέπει να επικεντρώσουμε καταρχάς σε προσπάθειές μας σε νομοθετικέ αλλαγέ. Αυτό απλό είναι. Όταν, όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, να διορθώσουμε κάτι, λέμε «Α, διορθώσουμε την νομοθεσία». Αυτό είναι εύκολο. Το θέμα είναι να κάνουμε κάποιες προτάσεις για δύο κυρίως θέματα, ούτως ώστε να αφαιρέσουμε κάποιες από τις ε, διαδικασίες που περιπλέκουν την απλουστευμένη χρήση επιλογών για το κόστος και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, που όμως είναι πολύ περίπλοκο θέμα. Αν θέλετε να κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις και τι θα συμπεριλαμβάνει η έκθεση πιο λεπτομερός. Εδώ έχω μαζί μου το γραμματέα της ομάδας υψηλού επίπεδου. Θέλω να σας πω ότι βασιζόμαστε στην ε, γνώση των μελών της ομάδας που έχουν επιλεγεί από διάφορους τομείς. και που ξέρουν πολύ καλά αυτά τα θέματα. Μπορώ να σας δώσω και τον κατάλογο διαφόρων οργανώσεων και της ε, οργάνωσης της Συνομοσπονδίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Έχουμε ακούσει γνωμοδοτήσεις, απόψεις από τις περιφέρειες, από το Eurocities. Όλα αυτά τα έχετε στη διάθεσή σας στην πλατφόρμα μας. Προσπαθήσαμε να ακούσουμε διάφορους φορείς και έχουμε ζητήσει συνεισφορές από όλους που έχουν να πούν οτιδήποτε πάνω σε αυτά τα θέματα. Για το ελεγκτικό συνέδριο. Στην πρώτη μας συνεδρίαση είχαμε και ένα μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Αλλά πάνω απ' όλα εμείς υπηρετούμε την Κομισιόν. Θα υποβάλουμε τις προτάσεις μας στην Κομισιόν. Θα έρθω σύντομα σε επαφή με την κυρία Γκρέσλερ από την ε, Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών για να συζητήσουμε για πιθανή συνεργασία με την Επιτροπή αυτή. Δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη πρόταση τι θα κάνουμε με αυτό τον όγκο πληροφοριών που έχουμε για το guidance. Η σύγχυση που υπάρχει οφείλεται στο ότι το λάθος ερμηνεύεται με πολιτικό τρόπο. Όλοι φοβούνται να κάνουν λάθη. Οι διαχειριστικές αρχές οι κρατικοί φορείς, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, αλλά και οι κομισιόν. Όλοι προσπαθούν να βρουν διευκρινήσεις, ερμηνείες, ε, τρόπους για να αποκλειστεί το λάθος. Εν συνεχεία, τι κάνουμε με αυτή τη διαδικασία. Επιβάλλουμε περισσότερους κανόνες, με περισσότερες λεπτομέρειες και αυξάνουμε την πιθανότητα έτσι για λάθος, για σφάλματα. Είναι τεράστιο θέμα και εξόχως πολιτικό όταν ζητούνται περισσότερες ε, επεξηγηματικά μνημόνια, ερμηνείες, εγκύκλοι από τα κράτη-μέλη, όταν τα κράτη-μέλη θέλουν να μάθουν περισσότερα, τότε πραγματικά εδώ πρέπει να παίξει το ρόλο του Κοινοβούλιο, να ακούσουμε τις προτάσεις σας, να συζητήσουμε αυτά τα μείζωνα θέματα μαζί σας, γιατί υπάρχουν δύο θέματα. Καταρχάς είναι αυτά που εύκολα μπορούμε να πετύχουμε, και από την άλλη κάποιες προτάσεις που αφορούν ε, γενικά α, τον τομέα αυτό πέρα από τη συγκεκριμένη περίοδο προγραμματισμού και που αφορούν και το θέμα της ήπιας νομοθεσίας. Αλλά αυτό συνδέεται και με το λεγόμενο gold plating που θα συζητήσουμε τον Ιούνιο. Την προσπάθεια των κρατών μελών, δηλαδή να ερμηνεύσουν ε, τους κανόνες, ή να τους κάνουν πιο περιοριστικούς, ε, ή να μειώσουν τις πιθανότητες ερμηνείας για να αποφύγουν το λάθος. Ξέρετε από, ότι υπάρχουν δύο μέρη. Από τη μία είναι ο δικαιούχο και από την άλλη είναι ο πληρωτή. Και οι πληρωτέ είναι πάντα πολύ ύποπτοι για τη χρήση των ευρωπαϊκών ε, κονδυλίων. Και αυτή η φυσική επιθυμία των πληρωτών να εξασφαλίσουμε χρηστή διαχείριση των κονδυλίων, πώς θα την παντρέψουμε με την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα λεφτά από τους δικαιούχους με πιο ευέλικτο τρόπο. Τεράστιο θέμα. Προσπαθούμε λοιπόν να απλουστεύσουμε κάποιο σύστημα χορηγήσεων για τον τομέα των ερευνών. Και υπήρξαν επικρίσεις από τους ίδιους τους ερευνητές οι οποίοι δεν θέλανε να έχουν τόσο μεγάλη ευκαμψία γιατί είχαν δυσκολία να καταλάβουν ποια ποιες δαπάνες ήταν επιλέξιμες για επιστροφή κόστους. Νομίζω λοιπόν ότι αυτές οι απλοποιημένες ε, διαδικασίες για την κοστολόγηση εμπλέκουν και τα θέματα των κρατικών επιδοτήσεων. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα. Ξέρουμε όλοι ότι δεν πρέπει οι κρατικές επιδοτήσεις να οδηγούν σε στρεβλώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο λοιπόν παρακολουθείται από πολύ κοντά. Για τις ε, διαμεθοριακές τώρα διαδικασίες. Το Interreg είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στο πρόγραμμά μας, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και εδώ υπάρχουν διαφορετικές ε, προσεγγίσεις σε διάφορες χώρες. Και εμείς συνεργαζόμαστε μαζί με την Κομισιόν, τον κύριο Τίμερμανς, μέσα στα πλαίσια της καλύτερης ρύθμισης και συνεργαζόμαστε σε αυτό το θέμα. Για τα επίπεδα λογιστικού ελέγχου και για τους μικρούς δικαιούχους και εδώ έχουμε κάποιες προτάσεις για να μειώσουμε τον έλεγχο για τους μικρούς δικαιούχους και τις μικρές χορηγήσεις και επιδοτήσεις. Να υπάρχουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι μονάχα και όχι εξονυχιστικοί έλεγχοι και πρέπει να εξετάσουμε και τις προτάσεις για κατόφλια ελέγχου. Δεν συζητήσαμε το θέμα της απορρόφησης των κονδυλίων των διαρθρωτικών πόρων. Γιατί δεν είναι μέσα στην εντολή μας βέβαια. Όπως έχουν πει όμω οι συνάδελφοι, οι έντιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και θέλουμε να κάνουμε κάτι για όλα αυτά γιατί εγώ μπορώ να αναφερθώ σε πολλές ομάδες υψηλού επίπεδου, ομάδες σοφών, που τις έχει φάει η μαρμάγκα της ιστορίας. Κανείς δεν τις θυμάται πια, παρά τις προτάσεις που έχουν καταθέσει. Και επομένως θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πολιτικές αποφάσεις, σε μιζόνες πολιτικές αποφάσεις. Πόσα προγράμματα χρειαζόμαστε. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία επικρίνουν την ευρωπαϊκή ε, γραφειοκρατία, αλλά όταν πρέπει να έχουν ένα πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν, δημιουργήσαν τέσσερα προγράμματα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να βοηθήσει να δημιουργηθεί κάποιος μηχανισμός για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προγραμμάτων. Το θέμα των κατευθυντηρίων γραμμών και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πολιτικό θέμα και ο λογιστικός έλεγχος και οι διάφορες, τα διάφορα επίπεδα ελέγχου δεν πρέπει να είναι υπερβολικά. Για την διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφορικής. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα για την πληροφορική και αυτό προτάθηκε. Αλλά η Κομισιόν θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τέτοιο σύστημα αλλά από τη στιγμή που θα γίνει η πρόσκληση ενδιαφέροντος μέχρι την ε, εφαρμογή του θα χρειαστούν δεκαετίες και δεν είναι ρεαλιστικό να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορούμε όμως να εναρμονίσουμε τα πρότυπα για την ε, πληροφορική που μπορούν να εξασφαλίσουν την ε, διαλειτουργικότητα. Όπως είναι και με τη Microsoft και την Apple. Και θυμάστε ότι πριν από 15 χρόνια υπήρχε τελείως τέλεια έλλειψη συμβατότητας. Τώρα όλα είναι συμβατά, υπάρχουν οι εμπειρογνώμονες της πληροφορικής οι οποίοι μπορούν να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά και να εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα. Και αν θέλετε να θέσετε κάποια πιο συγκεκριμένα... Ο Μάρη ίσως να μπορεί να σας πει κάτι πιο συγκεκριμένο, αν θέλετε. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Ε, έχουμε 7-8 ερωτήσεις ακόμα. Σαφίρ. Ένα λεπτό παρακαλώ συνάδελφοι να κάνετε τις ερωτήσεις σας για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ. Η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών θεωρούν ότι οι εκπρόσωποι των κρατών μελών δεν θα, πρέπει, δεν θα έπρεπε να είχαν αποκλειστεί από την ομάδα υψηλού επίπεδου που δημιουργήθηκε για να απλουστευθούν οι κανονισμοί για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πιστεύουμε ότι οι εκπρόσωποι των κρατών μελών είναι εκείνοι που ξέρουν τα ε, προβλήματα και τα στρεβλά του συστήματός τους και μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση. Σας ερωτώ, σχεδιάζετε και αν ναι με ποιο τρόπο να τους εμπλέξετε στη μελλοντική σας δουλειά για να συνεισφέρουν. Ευχαριστώ κυρία Μάλιτιτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε κύριε Κάλλας. Με χαρά σας υποδεχόμαστε στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το ποια θα είναι η τελική έκβαση. Κάθε φορά που συζητούμε για απλοποίηση φυσικά περιπλέκουμε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Δημιουργούμε νέε κατευθυντηρίε γραμμές, φορτώνουμε τη βάρκα γιατί θέλουμε να απλουστεύσουμε τα πράγματα και αυτό είναι πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι η απλοποίηση σημαίνει ότι κάνω τα πράγματα διαφορετικά με άλλο τρόπο πιο φιλικό προς το χρήστη. Δηλαδή ενδεχομένως να δημιουργήσουμε κάποια κέντρα γνώσης και αριστείας σε περιφερειακό επίπεδο και εκεί αυτά με τη σειρά τους θα υποστηρίζουν τον τελικό δικαιούχο για να είναι σε θέση να καταλαβαίνει όλες αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές και τους κανονισμούς. Και να μην χρειάζεται ο κάθε δικαιούχο να τα μαθαίνει όλα αυτά. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχουν κανόνε για τι κρατικέ ενισχύσει, το είπατε κι εσεί, που είναι τόσο περίπλοκοι, ώστε οι τελικοί δικαιούχοι πελαγώνουν και δεν μπορούν να τα βγάζουν πέρα. Αν δημιουργούσαμε τέτοια κέντρα αριστείας όμως και γνώση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένως να συνιστούσε αυτό κάποια πρόοδο. Ευχαριστώ ο κύριος Έθριτς. Για ένα λεπτό πάντα. Ευχαριστώ. Ε, ε, πω από δουλειά που σας ε, έτυχε, κλήρος που σας έχει πέσει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόβλημα έτσι κι αλλιώς οι κανόνες. 800 σελίδες είναι ένα εγχειρίδιο Εσεί το κάνετε αυτό γιατί είναι τόσο πολλέ οι δικαιοδοσίε οι νόμοι και οι Η απλούστευση γίνεται με περισσότερη συνοχή. Συνοχή μπορεί να επιτευχθεί μόνο ε, βέβαια με θυσία εθνική κυριαρχία και αυτή είναι η τραγωδία ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να τα πετύχει όλα αυτά χωρί να υπάρχουν Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη, πράγμα που ο κόσμο ακριβώ δεν θέλει. Και ερώτηση ε, και σας ε, εύχομαι καλή τύχη για την αναθεώρηση αυτού του εγχειριδίου από τι 800 Πόσε θα το πάτε, αν είναι κάτω από 750 είναι μεγάλη επιτυχία. Εσείς πώς το βλέπετε, πώς το εκτιμάτε από σελίδε. Ευχαριστώ κύριος Χέκμαν για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ τον κύριο Κάλλας το εξής. Εσείς τι πιστεύετε δεν θα πρέπει η ομάδα σας, αυτή η ομάδα υψηλού επίπεδου, να επικεντρωθεί μόνο στη λεγόμενη ήπια νομοθεσία που είναι κατευθυντήρες γραμμές, όχι οι κανονισμοί. Συμφωνώ ότι αυτό είναι το θέμα και εκεί ε, είναι το κρίσιμο. Έχουμε κατευθυντήριες γραμμές ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε κανονισμούς στα κράτη-μέλη. Έχουμε προσανατολισμούς στη συνέχεια στα διαφορά ΕΣΠΑ, τα κρατικά και έχουμε ε, και κατευθυντήριες γραμμές εγχειρίδια που εξειδικεύουν ε, το εκάστοτε επιχειρησιακό σχέδιο. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές λοιπόν και οι προσανατολισμοί, πώς να το πω, είναι ένας τεράστιος όγκος που χρησιμεύει μόνο ε, για ενημέρωση, όπως είναι αυτές οι ενημερωτικές πινακίδες που βλέπετε στα έργα, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που χρειάζεται είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και των διαρθρωτικών ταμείων. Αν θέλουμε να τα απλοποιήσουμε όλα, θα χάσουμε. Δεν μπορούμε με μία προσπάθεια. Ε, ας περιοριστούμε στην ήπια νομοθεσία, στις κατευθυντήριες γραμμές και μόνο. Και θα πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση χρησιμοποιώντας την κοινή λογική στη διοίκηση και στις διαχειριστικές αρχές. Τα πάντα είναι θέμα εμπιστοσύνης άλλωστε. Πόσο πιθανό είναι να πριτανεύσει η κοινή λογική. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπρέσσο. Πολύ σύντομα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Να σας πω τι πιστεύω εγώ. Ο μόνος τρόπος για να πλουστεύσουμε πραγματικά είναι να έχουμε ένα άτομο που κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας είναι επιφορτισμένο και είναι το, η δουλειά του να μειώσει δραστικά τις α, ε, προτινόμενες ρυθμίσεις. Τον αριθμό τους δηλαδή. Δηλαδή, να μειώσει τον αριθμό των σελίδων, ας πούμε αν ας πούμε έχουμε 40 σελίδες αρχικά, να έχει το καθήκον να τις μειώσει σε 10. Και με προτάσεις και διάλογο μεταξύ σας τελικά καταφέρετε να το πετύχετε. Η βασική αρχή θα είναι ότι να μην, ζητάνε, ε, να μην ζητούνται πληροφορίες άχρηστες που δεν χρησιμοποιούνται και δεν έχουν νόημα για την νομοθετική διαδικασία. Δηλαδή, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν γίνεται μια επαλήθευση, οι περισσότερε είναι άχρηστε. Δεύτερον, η αρχή τη ε, ευθύνη. θα πρέπει να έχουμε την αρχή της ε, ευθύνης, αυτός που παρουσιάζει το, το πρόγραμμα, δηλαδή, να έχει αυτή την ευθύνη. Και εν συνεχεία, αν εγώ έχω παρουσιάσει ένα πρόγραμμα και έχω πάρει λεφτά, ε, θα πρέπει να δείξω αποτελέσματα. Αυτό μετράει. Όχι το να έχω ε, γεμίσει σελίδες και δελτία, ας πούμε, εκατοντάδες από αυτά. Και κάτι άλλο. Έχουμε εγκρίνει εμεί στο Κοινοβούλιο ε, ένα κείμενο για όλα τα διευθυντικά ταμεία. Εν συνεχεία είχαμε τέσσερις κανονισμούς, ένα ένα ταμείο. Δηλαδή, αγνοήσαμε εντελώ στην αρχή ότι θα πρέπει να έχουμε μία, ε, δηλαδή μία, ένα κανονισμό, ε, μια και τα ταμεία έχουν πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά. Και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Ε, αν μπορούμε να έχουμε ένα κανονισμό, γιατί να έχουμε τέσσερι. Γιατί αυτό παραβιάζει ε, την αρχή τη απλούστευσης. Και όταν φτάσουμε στα τέσσερα, μετά θα πάμε στα πέντε κείμενα. Και τελικά οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ιδέα ποιο κανονισμό ισχύει, γιατί δεν έχουν και τόσε διαφορέ μεταξύ του. Ευχαριστώ κύριε Τσέλερ. Ε, σύντομα σα παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να καλωσορίσω και τον επίτροπο κύριο Κάλλα και να του ευχηθώ μεγάλη καλή επιτυχία γιατί δεν είναι τόσο εύκολο το έργο του. Μικρόφωνο. Α, είναι μακριά, ναι. Λοιπόν, έλεγα, κύριε Κάλλα, καλή επιτυχία δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο σας. Τώρα κοιτάξτε, λείπει ένας πάρα πολύ σημαντικός φορέας και θέλω να συμφωνήσω με την κυρία Τόμασιτ και να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε. Σε ό,τι αφορά την νομοθετική διαδικασία, εδώ είμαστε στη συναπόφαση. Έχει λόγο δηλαδή και το Συμβούλιο και για την υλοποίηση των προγραμμάτων και την εκτέλεσή τους και τις εταιρικέ ε, σχέσεις. Είμαστε στη ε, συνδιαχείριση και είναι αρμόδια τα κράτη-μέλη και πάλι δηλαδή τα μέλη του Συμβουλίου. Ε, τώρα θα πρέπει να έχουμε λόγο κι εμείς. Όποιος έχει ζήσει τριμερή διάλογο γνωρίζει ότι, όπως λέμε στη Γερμανία, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι διότι έχουμε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τροπολογίες στο Κοινοβούλιο και μετά καμιά φορά χρειάζονται μήνε για να μην πω και χρόνια, που αλλάζουν διάφορε προεδρίε και τώρα κάθε χώρα ε, έχει τον πόνο τη και τι απαιτήσει τη και ε, φτάνουμε στι 280 σελίδε μόνο για ένα κανονισμό. Μετά πάει αυτό στις ομάδες εργασίας για την εκτέλεση και εκεί ε, συνεδριάζουν οι υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι είναι πάντα πάρα πολύ σχολαστικοί και έχουν ε, ρυθμίσεις θέλουν να έχουν πάρα πολύ λεπτομερείς εντολές και υποδείξεις για να έχουν πιο εύκολη δουλειά. Και στο βαθμό που είναι έμπειροι, ε, που ξέρουν περί τίνος πρόκειται και ξέρουν να το χειριστούν. Όταν η διοίκηση έχει συνέχεια δεν υπάρχουν δυσκολίες. Εκεί που αλλάζουν συνεχώς οι υπάλληλοι της διοίκησης έχουμε προβλήματα. Γιατί δεν ξέρουν να εφαρμόζουν αυτά τα πράγματα και τις δύσκολες και περίπλοκες διαδικασίες πρέπει να τις μαθαίνουν κάθε φορά από την αρχή. Και ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας είναι οι τελικοί δικαιούχοι που διαχειρίζονται τα προγράμματα που τους έρχεται στο κεφάλι ένας κικαιώνας ρυθμίσεων και δεν έχουμε φτάσει σε 880 σελίδες στο κατευθυντήριο γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους εμβούλιο που τους έχουν διαπραγματευτεί, αλλά έρχεται να προσκεφτεί και η συνδιαχείριση. Χαιρετίσματα, γιατί έρχονται και οι εθνικές ρυθμίσεις επιπλέον. Και όποιος έχει ακόμα το κουράγιο στα πλαίσια της συνοχής να υλοποιήσει ένα έργο, δεν μπορώ παρά να το συγχαρώ και να του βγάλω το καπέλο. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τις διαδικασίες και τις μεθόδους που θεσπίζουμε, αυτό να συζητήσουμε και μήπως εκεί χρειάζεται και χωράει περισσότερη διαφάνεια. Και να είμαστε και πιο προσιλωμένοι στο στόχο μας. Και ως μέλος Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα ήθελα να πω ότι στόχος της Επιτροπής μας δεν είναι να έχουμε ε, ένα τεράστιο κανονισμό και ρυθμίσεις που ε, ήδη ενέχει ε, τα σφάλματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου να πιάνουν τόπο με στοχοπροσύλωση, με διαδικασίες αποτελεσματικές και να είναι όλα αυτά εύστοχα και με επιμέλεια και με ε, προσοχή και με αποτελεσματικότητα να γίνεται η διαχείριση. Εάν επιτευχθούν όλα αυτά, είναι ικανοποιημένη και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και δεν χρειαζόμαστε τέτοια μεγαλειώδη ε, κανονισμούς και ρυθμίσεις. Ο κύριος Νοβάκοφ είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ένα λεπτό είχα παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρο. Χαίρομαι που κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αναφέρθηκε και το θέμα του ψηφίσματος που εγώ θέλησα να ξεκινήσω πέρσι. Είχα την τελευταία εβδομάδα επαφές με δικιούχους στη χώρα μου που έχουν επιβεβαιώσει τους φόρους μου σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχής. Γιατί εδώ στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου φαίνονται μηχανισμοί ότι είναι αποδεκτοί. Όταν φτάσει όμως στο εθνικό επίπεδο υπάρχει το gold plating, η προσθήκη κανόνων που ακόμα περισσότερο ε, επιβαρύνουν το δικαίωχο. Και όταν φτάσουμε στο τοπικό επίπεδο, οι τοπικές αρχές κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση για το δικαιούχο γιατί έχουν επιπλέον ε, επιβολές που ζητούν από το δικαιούχο. Λοιπόν, αρκετά συζητήσαμε, για το πρόβλημα, συζητήσαμε το πρόβλημα, θα πρέπει να δούμε τώρα ποιες είναι οι λύσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι ήδη με την ενδιάμεση αναθεώρηση το 2018. Δεν λέω ότι μπορούμε να λύσουμε όλο το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον κάποιες τροποποίησεις στους κανονισμούς. Σε κάποιους τομείς λοιπόν θα ήταν χρήσιμο να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποιες τέτοιες λύσεις και να τις συζητήσουμε. Η παρακολούθηση των στόχων της συνοχής και τα θέματα των δημοσίων προμηθειών. Και αυτό μήπως θα μπορούσε να είναι ένα τμήμα της λύσης. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Όπως βλέπετε, κύριε Κάλλας, πολλές είναι οι ερωτήσεις και μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση για πολλές ώρες. Στο μέλλον τώρα σας δίνω όμως ένα πολύ σύντομο διάστημα για να απαντήσετε μονάχα σε αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, τα κράτη-μέλη συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα εργασίας Δύο υφυπουργού και πέντε διευθυντέ υπουργείων από τα κράτη-μέλη συμμετέχουν σε αυτήν την διαδικασία. Συμμετέχουν λοιπόν τα κράτη-μέλη χωρίς καμία αμφιβολία. Όπως είπε ο κύριο Τσέλερ βέβαια, εμπλέκεται το θέμα των φορολογουμένων και της ανησυχία των φορολογουμένων να χρησιμοποιηθούν σωστά τα χρήματα. Γι' αυτό υπάρχουν και τόσα πολλά θέματα τα οποία τίθενται σε σχέση με τις πρόσθετες κατευθυντήρες γραμμές και τις ερμηνείες τους. Πώς θα βγούμε από αυτό τον κικαιώνα είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Δεν θέλουμε βέβαια να οδηγηθούμε σε περαιτέρω κατευθυντήρες γραμμές για περαιτέρω απλοποίηση που θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερο χαρτοβασίλειο. Και φυσικά εδώ εμπλέκεται η πολιτική ευθύνη της ομάδας μας που θα πρέπει να βρει τρόπους να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα για τον αριθμό των σελίδων. Δεν μπορώ να σας πω σήμερα. Όταν έχουμε όμως κάποια αποτελέσματα και περιορίσουμε το μήκος στον κανονισμό, αυτό θα είναι ε, χρήσιμο. Και για τα εύκολα που είπατε, η τελική μας έκθεση δεν θα είναι το 2018, θα πρέπει πρώτα να καταλήξουμε σε κάποια πορίσματα τα οποία θα σας παρουσιάσουμε. Και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να ανταποκριθούμε για να δούμε τι μπορεί να γίνει σε μικρά πράγματα και ελπίζω ότι η Κομισιόν θα τα πρώτη σε αυτά τα θέματα. Και οι νομοθετικές προτάσεις. Άμα κάνουμε νομοθετικές προτάσεις, θα χρειαστεί περισσότερος καιρός. Για τις διαδικασίες. Οι κατευθυντές γραμμές αφορούν τις διαδικασίες ιδίως. Εκεί είναι τα πιο μεγάλα προβληματικά θέματα. Εκεί είναι που οι ελεγκτές βρίσκουν τα περισσότερα σφάλματα, κυρίως στις διαδικασίες όταν αντιμετώπιζα αυτό το θέμα. Αυτό είχα καταλάβει. Υπήρξαν λοιπόν αυτά τα σφάλματα στην διαδικασία τα οποία ε, μπορούσαν να διορθωθούν στο τέλος αλλά η ζημιά είχε γίνει. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολιτικά πολύ σημαντικά να τα επιλύσουμε και δημιουργούν και καχυποψία. το να έχετε ένα άτομο το οποίο είναι αρμόδιο για την απλοποίηση. Η Κομισιόν έχει βάλει τον κύριο Τίμερμανς ως αρμόδιο για την καλύτερη νομοθεσία. Ο κύριος Τίμερμανς είναι ο κύριος υπεύθυνο για τα θέματα απλοποίησης σε πολιτικό επίπεδο. Δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει, αλλά η Κομισιόν νομίζω έχει αρχίσει να είναι πιο κριτική στην ε, αντιμετώπιση νέων κανονισμών και νέων προτάσεων. Και επομένως αυτή είναι η κατευθυντή διαγραμμή της Κομισιόν. Και τέθηκε το ερώτημα από εσά και έχει τέθει και στην ομάδα εμπειρογνωμόνων το θέμα για την βασική οντολογική έννοια των κατευθυντηριών γραμμών και της αύξησής του από τα κράτη-μέλη, το λεγόμενο gold plating, την χρυσοπίκυλση. Νομίζω ότι όπως λένε πάρα πολύ όλα αυτά είναι αδύνατο να τύχουν διαχείρισης. Θα πρέπει να υπάρξει κάποιο ξεκαθάρισμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ λέει και η πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Κάλλας. Χρειάζομαστε μια περαιτέρω συζήτηση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις ανταλλαγές απόψεών μας με την ομάδα σας και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όπως βλέπετε να ακούσουμε τις απόψεις σας για τα θέματα αυτά. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι. Και τώρα ερχόμαστε στον χρόνο ψηφοφοριών. Έχετε τις κάρτες σας όλοι ελπίζω αν χρειαστεί να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, βεβαίως. Okay, before, before we begin... Uh, Πρώτον ξεκινήσουμε. Μου είπε η γραμματεία ότι περισσεύουν κάποιοι από την ομάδα των φιλελευθέρων. Έχουμε τέσσερις έδρες. Ναι, ναι, εντάξει, θα μείνω και ο Στάκουλα. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινούμε με την έκθεση, με την έκθεση της κυρίας Τόματσιτς. Νέες νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 2014-2020, ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και οδηγούμενες από τις τοπικές κοινότητες, τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Η συγγήτριά μας έχει παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσή τη τον Δεκέμβριο με χρήτη καταληκτική Προθεσμοί είχαμε πάρει 171 τροπολογίες και η Επιτροπή Απασχόλησης έχει προετοιμάσει και αυτή μια γνωμοδότηση και η συγγήτρια προτείνει μια σειρά από συμβαστικέ τροπολογίε. Θέλετε να λάβετε το λόγο, κυρία Τόμασιτ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας και για τις προτάσεις σας και για τις τροπολογίες σας. Το κοινό μας εργασί, έργο έχει οδηγήσει σε μια πολύ καλή έκθεση και σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας. Καλά. Μπορούμε να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία επομένως. Ξεκινούμε με την τροπολογία συμβασμού 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχέ. Νόμιζα ότι απορρίπτεται αλλά κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απέριπτε. Τροπολογία 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Για την 97 ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε πράγματι. 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική εννέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόλ 4. Έμπλ 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έμπλ 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλ 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά ποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 118 υπέρ κατά αποχές αθετείται έμπλ 5 υπέρ κατά εποχές Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Την Apple 5. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 119 υπέρ. Κατά. Υποχές. Απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, εποχές, υιοθετείται. Συμβασμός 11 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Έμπλ 11 υπέρ, κατά, εποχές υιοθετείται. Τροπολογία 124 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 12 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 136, τροπολογία 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 13. Λάβαμε το εξής έτοιμα. Από το ΕΛΚ ε, έτοιμα για χωριστή ψηφοφορία, ψηφοφορία κατά τμήματα, σε τέσσερα τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα του Συμβασμού 13. Υπέρ κατά αποχές Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα του 13 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. Σημασμός 13, τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 13, τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στο συμβασμό 14 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Τροπολογία 147, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 148 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 149 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά εποχές ελέγχουμε χρονικά την 155 πέρας υιοθετείτε 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Συμβιβασμός 15 υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. 163 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές. Φαίνεται ότι υιοθετείται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 167 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβιβασμός 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 171 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε Τροπολογία 1 υπέρ κατά εποχές υιοθετείτε 2 υπέρ κατά εποχές υιοθετείτε 3 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά εποχές υιοθετείτε 6 υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε 9 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε μάλλον. 9 ψηφίσαμε μόλις τώρα, στο 17, υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 13 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά εποχές υιοθετείται 16 υπέρ κατά εποχές υιοθετείται 17 υπέρ κατά εποχές υιοθετείται 18 υπέρ κατά εποχές υιοθετείται 19 υπέρ καταπίπτει 19 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα θα πάμε στην τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 28 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η συμβαστική υπέρ 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπέρ 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 34 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Και τώρα η τελική ψηφοφορία για το σύνορο του ψηφίσματος ηλεκτρονικά παρακαλώ αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια. Now with our next... Συνεχίζουμε. Έχουμε την επόμενη ψηφοφορία τώρα γνωμοδότηση για την απαλλαγή του 2014 Γενικός Προπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συγκήτρια είναι η κυρία Μάλετιτς. Θέλετε να πείτε τίποτα? Όχι. Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε μέσω στην ψηφοφορία. Πάμε λοιπόν. Συμβαστική υπαριθμόν 1. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 2 ψήφι περ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική υπαριθμό 2, έτσι δεν είναι, ψήφι περ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 22 υπέρ, κατά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 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίψετε. Η τροπολογία υπάρχει 58 υπέρ, κατά, αποχές, αυτό θέλει έλεγχο. Την 58 ελέγχουμε ηλεκτρονικά τώρα, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα θα πάμε στο σύνολο της γνωμοδότησης, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίθηκε η γνωμοδότησή μας. Συγχαρητήρια, κυρία Μάλετη. We continue. Συνεχίζουμε. Στην... στην γνωμοδότηση για τον συντονισμό, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Επισκόψη Ετήσιας Ανάπτυξης 2016. Εγώ ήμουν εισηγήτρια. Ξεκινάμε λοιπόν με τη συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές Εγκρίντ. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές Εγκρίντ. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτονται. 43 εκπίπτει. Σαράντα με προφορική τροποποίηση. Υπάρχει αντίληση για την προφορική τροποποίηση. Όχι. 44 λοιπόν με την προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν η γνωμοδότησή μας. Ευχαριστώ. Η γνωμοδότηση τώρα του κυρίου Κοτσολίνο για την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική για μια ολιστική προσέγγιση στη μετανάστευση. Κύριε Κοτσολίνο, θέλετε να πείτε κάτι. Καλά. Ψηφοφορία. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για τη συμβαστική 2. Ηλεκτρικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Συγγνώμη, συγγνώμη, έκανα... Ήταν φανερό, δεν χρειάζεται να έλεγχο. 29-8. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ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 The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση αυτή και σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια κύριε Κοτσολίνο μου. Σας ευχαριστώ. Ολόκληρη Επιτροπή. Κάναμε καλή δουλειά. Έχω δύο σχόλια ακόμα όμως. Οι συντονιστές συνεδρίασαν εκτές και έλαβαν κάποιες αποφάσεις οι οποίες σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικώς με mail. Δέχεστε, εγκρίνετε τις αποφάσεις των συντονιστών, μάλιστα, ευχαριστώ. Διάφορα. Έχει κανείς κανένα διάφορο, καμιά ερώτηση. Όχι. Να σας θυμίσω μόνο την προσεχή μας συνεδρίαση. Είναι τη Δετάρτη 16 Μαρτίου το απόγευμα και 17 Μαρτίου μέρα Πέμπτη το πρωί. Ευχαριστώ τους Δερμηνείς και οι Δερμηνείς ευχαριστούν. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Λήξη συνεδρίας.